Uh, okay, colleagues, I think we'll make a start. It's... Uh, Καλημέρα συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Είναι 9.35 και 35 και αντικαθιστώ την πρόεδρο σήμερα το πρωί, διότι προετοιμάζεται και μετά θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για τις τριμερείς συνομιλίες. Επομένως σήμερα το πρωί θα είμαι εδώ εγώ και θα δούμε αν θα γυρίσει για το απόγευμα. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ζητήσω είναι να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αλλαγές, νομίζω ότι μπορούμε να θεωρούμε, θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται. Έχω κάποιες ανακοινώσεις εξ ονόματος Πρόεδρου. Ξέρω ότι σας έχει ανησυχήσει ο αριθμός των έκτακτων συνεδριάσεων που έγιναν σε Στρασβούργο και εγώ θεωρώ ότι είναι επιπρόσθετο το άχθος για το πρόγραμμα των Ευρωβουλευτών και δυστυχώς ε, το πρόγραμμα που έχουμε στην Επιτροπή μας ε, σημαίνει ότι προς το παρόν και σε αυτό συμφώνησαν και οι συντονιστές ε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να παρακολουθούμε τα θέματα τα οποία μας έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς το παρόν λοιπόν θα γίνονται ακόμα έκτακτες συνεδριάσεις στο Αεροσβούργο. Επίσης θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση για την εκτύπωση των εγγράφων της Επιτροπής. Θα έχετε προσθέσει, προσέξει από τον μεγάλο αριθμό εγγράφων που έχετε στα έδρανά σας ε, ότι ίσω καταναλώνουμε λίγο παραπάνω χαρτί εδώ στην Επιτροπή και διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή έχει εκτυπώσει πολλές φορές τα ίδια έγγραφα. Αυτή τη στιγμή τα εκτυπώνουμε τρεις φορές τα ίδια έγγραφα. Φαίνεται ότι δεν κάνουμε τίποτα καλό για το περιβάλλον ως Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε και αυτό υποστηρίχθηκε από όλους ότι θα εκτυπώνονται τα έγγραφα μία φορά και από εκεί και πέρα θα είναι διαθέσιμα ε, στις ιστοσελίδες της Επιτροπής ε, ε, θα έχετε πρόσβαση λοιπόν στις ιστοσελίδες και αν κάποιος χρειάζεται επιπλέον έγγραφα μπορείτε κάλλιστα να ζητήσετε εκτύπωση από την υπηρεσία τεκμηρίωσης. Δεν παραβιάζετε δηλαδή το δικαίωμά σας να έχετε τα έγγραφα, απλώς είναι τεράστια σπατάλη να τα τυπώνουμε τρεις φορές για όλους στη διάρκεια της των συνεδριάσεων των επιτροπών. Θα ήθελα τώρα να κάνουμε ένα διόδρομο στην οδηγία προσπέκτους όπως υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι θα το λάβατε αυτό. Βάσει του άρθρου 216 του κανονισμού ε, θα εγκρίνουμε αυτό το διορθωτικό έγγραφο. Να σας ε, επισημάνω ότι εδώ απλώς ε, διορθώνονται οι πράξεις στη κατεξουσιοδότηση και εισάγεται μία μικρή παράγραφος η οποία υπήρξε αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αυτή η νέα παράγραφος, άρθρο 3, ε, συγγνώμη, παράγραφος 3 άρθρο 8 εγκρίθηκε ε, παραμένει στο τελικό κείμενο. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, εγκρίνεται και θα ανακοινωθεί στην επόμενη συνεδρία της Ομιλομέλειας. Μία τελευταία ανακοίνωση το ψήφισμα για για τα μη ανταγωνιστικά ορυχεία θα περάσει ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό το οποίο ε, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά ε, την Επιτουσουσίας Επιτροπή. Η Επιτουσουσίας Επιτροπή είναι η Επιτροπή μας και εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε τι ε, πορεία θα ακολουθήσουμε. Αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε έκθεση βάσει του κανόνα 48 για την περίπτωση των μη ανταγωνιστικών ανθρακοριχείων ε, Ούτω ή άλλω είναι στο πρόγραμμά μας, ετοιμάζει κάτι ο εισηγητή, ο κύριος Ραπ Κάι και επομένω μπορούμε να καταθέσουμε τη μετροπολογία σε αυτή την έκθεση μέχρι τις 26 Οκτωβρίου και μετά ε, θα το ψηφίσουμε στις 9 Νοεμβρίου. Οι συντονιστές ε, σωστά λοιπόν αποφάσισαν ότι το ψήφισμα δεν θα προχωρήσει και ε, οι συντάκτες του ψηφίσματος θα ενημερωθούν ότι υπάρχει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή. Αν υπάρχουν σχόλια επί των ανακοινώσεων, να σα ακούσω. αλλιώ νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο πρώτο θέμα τη ημερήσια διάταξη στο σημείο 3, φορολογία και ανάπτυξη, συνεργασία με τι αναπτυσσόμενες χώρε για την πρόθεση της χρήσης κυβέρνηση στο φορολογικό τομέα. Η συντάκτρια τη νομοδότηση είναι εδώ, να τη δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όπως uh, είδαμε πρόκειται για θέμα καλής διακυβέρνησης, το οποίο έχει τρεις πτυχές. Καταρχήν, να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά καλύτερη φορολογία, ανάπτυξη καλύτερου φορολογικού συστήματος. Δεύτερον, το θέμα των διασυνοριακών πολυεθνικών εταιριών, τη διαφάνειας όσον αφορά τα συστήματα φοροαποφυγής τους και τρίτον τις ε, διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ε, φορολογικών συστημάτων και της ε, φορολογίας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εγώ πιστεύω ότι Η τροπολογία 9 της ομάδας μου μπορεί να θεωρήσει ότι η τροπολογία 9 δεν ε, μπορεί να γίνει δεκτή, 16 τροπολογίες μπορούν να γίνουν δεκτές. Όσον αφορά τις διασυνοριακές ε, επιχειρήσεις, Θέλουμε να καλύψουμε το θέμα αυτό με μια συμβιβαστική τροπολογία ή με συμβαστικές τροπολογίες. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε συμφωνήσει. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των χωρών θα πρέπει να υπάρξει μια αναχώρα παρουσίαση, έκθεση. Η οδηγία για την διαφάνεια θα πρέπει επίσης να τύχη εξυγχρονισμού. Εδώ καλύπτουμε τα θέματα των, ε, της διαφάνειας με τις εταιρείε με έναν ομοιόμορφο τρόπο. Θέλουμε διαφάνεια και όσον αφορά τις οικονομικές πληροφορίες που δίνουν οι πολυεθνικές εταιρείε που παρέχουν και επίσης θα πρέπει να καλυφθεί το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου. Θα σε ευχαριστώ. Οι συγητές, οι σκιώδεις δεν είναι εδώ. Υπάρχουν προβλήματα πλήσεων από ό,τι μου είπανε. Ο κύριος Σνίτ από την ομάδα των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Είναι εξαιρετική η έκθεσή της και δύο τροπολογίες ελάσσων σημασίας, οποίες θέλω να πω ότι έχουν γίνει δεκτές, αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Το θέμα των ε, χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών και της φορολόγησης τους. Αυτό μπορεί να είναι ένα θέμα προβληματικό. Στην έκθεση Μπέρες υπήρξε μια προφορική τροπολογία των πρασίνων, την οποία εμείς ε, την απορρίψαμε. Και θέλουμε να υπάρξει μια πολύ πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος αυτού. Αλλά τελικά, στην τελική ψηφοφορία, όντως υπάρχει αυτό που αναφέρεται εδώ στην τροπολογία 9, διότι χάσαμε την ψηφοφορία. Πιστεύω λοιπόν ότι για όλους μας θα ήταν χρήσιμο να ξέραμε τι είναι το αποτέλεσμα τελικά. Διότι το θέμα αυτό αποκτά όλο και περισσότερη σημασία. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπατε, συμφωνώ με την εισηγήτρια, αλλά δεν ξέρω μήπως θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με αυτό που εδώ προτείνει η Επιτροπή και να έχουμε μια καλύτερη θέση του Κοινοβουλίου. Θέλετε να απαντήσετε στο τέλος, να ακούσουμε όλες τις παρατηρήσεις. Η κυρία Ποδηματά είναι αυτή η οποία θα οργανώσει και την ακρόαση στις 10 Ιανουαρίου. Ουσιαστικά λοιπόν η εργασία γίνεται από πολλές πλευρές, διότι δεν είναι μόνο το θέμα των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι πρέπει να το δούμε με πιο συνολικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. το μήνυμά μου είναι από τον ε, Δ. Κανάλ και θα ήθελα να το διαβάσω. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την πάρα πολύ ισορροπημένη προσέγγιση της όσον αφορά την ανάπτυξη και τη φορολογία. Ζητούμε μια ρύθμιση, περισσότερη διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι καθοριστική για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο οι επιχειρηματίες θα μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στις επιχειρήσεις τους. Βεβαίως μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και η ανάπτυξη του δημόσιου τομέα, όχι όμως εις βάρο του ιδιωτικού τομέα. Χρειάζεται λοιπόν ένα προοδευτικό σύστημα φορολογία για τις αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι το οποίο δεν θα επηρεάσει τα χαμηλά εισοδήματα. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν τέτοιες φορολογικές πολιτικές να αναγνωρίζουμε ότι διευρύνεται η φορολογική βάση προωθώντας τους στόχους ανάπτυξης. Την ίδια ώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν οι κατευθυντήρες γραμμές του ΟΣΑ που βασίζονται στην αναχώρα παρουσίαση προτάσεων και οι αρμόδιες φορολογικές αρχές θα πρέπει να έχουν τον τρόπο να επιλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες και οι επιχειρηματίε θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν τον τόπο στον οποίο θα δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις τους. Πρόεδρος, βλέπω ότι οι σκιώδεις δεν είναι παρόντες και θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να πω στον κύριο Σμιτ, έχει δίκιο. Τροπολογία 9 λέει ακριβώς το ίδιο με αυτό που ψηφίσαμε στην Ολομέλεια όσον αφορά τις ε, φορολογήσεις των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Είναι μια ισορροπημένη διατύπωση και πιστεύω ότι πρέπει εδώ να το συζητήσουμε. Είναι όμως ε, ορθό το ότι η ομάδα μας δεν είναι υπέρ. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση παρόλα αυτά, γιατί καλό θα ήταν και στις δύο εκθέσεις η διατύπωση να είναι κοινή. Πρόεδρος, προοδεύει νομίζω η εργασία μας και θα πρέπει εδώ να φανεί καθαρά ποια είναι η άποψη του Κοινοβουλίου, αφού το θέμα αυτό συζητήθηκε και στην Ολομέλεια και αφού υπάρχουν παρόμοιες προτάσεις με σε άλλες εκθέσεις, θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση. would you Θέλετε, Νιόκ, να πάρετε το λόγο. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα με τις πτήσεις και όλος και όδης δεν έχει φτάσει. 9 Νοεμβρίου, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξει η ψηφοφορία 9 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή μας και τον Ιανουάριο στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ και μπορούμε τώρα να περάσουμε στην έκθεση του κυρίου Κάζα. Είναι το σημείο 4, κοινό σύστημα για την προστιθέμενη αξία με την υποχρέωση για τη διάρκεια υποχρεωτική εφαρμογή. Ευχαριστώ. Καλημέρα σα, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Το σύστημα, όπω είπαμε, δεν ε, είναι το καταλληλότερο και χρειάζεται οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί. Τα ζητήματα που τίθενται εδώ είναι περίπλοκα και πρέπει να γίνουν αλλαγές προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο δρόμο να προχωρήσουμε. Ω Κοινοβούλιο πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει κατά τρόπο αποτελεσματικό και έγκαιρο. Η Επιτροπή μας διαβεβαίωσε ότι θα δημοσιευθεί πράσινη βίβλος, η οποία θα δώσει περισσότερες αφορμές για συζήτηση. Τώρα οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί πρόκειται να ενισχύσουν τον όλο διάλογο που θα έχουμε και χαίρομαι που δεν πέσαμε στον πειρασμό να κάνουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις σε τόσο προκαταρκτικό στάδιο Δεδομένης της πολυπλοκότητας του ζητήματος, καθώς και της πολιτικής του σημασίας, νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη συζήτηση προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική η εσωτερική αγορά και να βεβαιωθούμε ότι το σύστημα μπορεί να καταπολεμά την απάτη. Γι' αυτό το λόγο δεν έχω αντιρρήσει στην τροπολογία 3 και 4 και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να θεσπίσουμε ένα νέο σύστημα, πράγμα που ελπίζουμε να είναι εφικτό όσο δυνατόν συντομότερα. Για αυτού του λόγους δεν έχω αντιρρήσεις στι τροπολογίε ε, του κ. Τάλια. Δεν είναι αμφιλεγόμενη η έκθεση, οπότε δεν έχω και άλλα σχόλια. Μάλιστα, πολύ κατανοητό. Είναι σκιώδη τώρα, ο κύριος Τάλερ. Για του σοσιαλιστές και δημοκρατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριο Κάζα είπε ότι δεν αμφιλεγόμενη η έκθεση. Εγώ στηρίζω τη δουλειά του και τον ευχαριστώ για όσα έχει κάνει. Πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο να στηρίξουμε το σύστημα του κατώτατου κανονικού συντελεστή του 15% για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα ώστε να εξασφαλιστεί νομική ασφάλεια. Όμως, εν τέλει θα χρειαστεί περαιτέρω αναθεώρηση. Ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η ενιαία αγορά θα πρέπει να διέπεται από κατευθυντήριε γραμμέ σε σχέση με αυτό το σύστημα. Το να έχουμε ένα οριστικό καθεστώ ε, πριν το τέλο τη παράταση, 21 Δεκεμβρίου 2015, είναι κάτι που θα πρέπει να το ευνοήσουμε. Υπάρχουν νέες οικονομικές πραγματικότητες, νέες τάσεις στην ε, φοροδιαφυγή και όλα, αυτά απαιτούν από μας να προσαρμόσουμε αναλόγως την νομοθεσία. Περιμένουμε λοιπόν από την Επιτροπή να επανεκτιμήσει αυτέ τι νέε πραγματικότητε και να προτείνει μια νέα στρατηγική για τον ΦΠΑ όσο δυνατόν συντομότερα. Και ή δυνατόν πριν το τέλο τη περίοδου που αυτή τη στιγμή προβλέπουμε να παρατείνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σμιτ για του φιλελεύθερου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Η τροπολογία σα κύριε Κάζα Μάλλον, η πρότασή σας για τις τροπολογίες είναι να είμαστε συντομότεροι. Μιλάτε για το 2013. Η πρόταση αρχικά είναι το 2015. Και εσείς είπατε ότι συμφωνείτε με τον κύριο Τάιλερ. Αλλάζετε δηλαδή, μεταλλάξετε τη τάση σας. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δράσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Γι' αυτό θα συμφωνήσω με την προηγούμενη σας πρόταση για το 2013. Δεν είναι και τόσο σημαντικό το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι το σύστημα ως έχει δεν είναι το καταλληλότερο, οπότε όσο πιο, δυνατο, πιο γρήγορα δράσουμε τόσο καλύτερα θα είναι για τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση σας ακολουθώ κύριε Κάζα. Πρόεδρος, δεν... Θα απαντήσει βέβαια ο κύριος Κάζα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. Ο κύριος Τάλερ είπε πριν το 2015. να αφήσω τον κύριο Κάζα ίσως να απαντήσει, αλλά προηγουμένως θα αφήσουμε τον κύριο Φόξ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι σχετικά απλή η πρόταση στόχο είναι να καταπολεμηθεί η απάτη και τα κράτη-μέλη συμφωνούν ότι το κατώτατο όριο του 15% πρέπει να παραταθεί το 2015 και το Κοινοβούλιο στηρίζει αυτή την ε, απόφαση. Επίση, θα συμφωνήσουμε με τι τροπολογίε του εισηγητή του κυρίου Κάζα. Τον ευχαριστώ για τη δουλειά του και να πω ότι στηρίζω τι τροπολογίε που πρότειναν ο κύριο Σμιτ κυρία Ασάγια. Είναι πολύτιμε για την έκθεση. Απλώ δεν ξέρω ακόμα αν θα στηρίξω τι τροπολογίε 5 και 6 του κυρίου Τάλ. Συμφωνούμε ότι η πράσινη βιβλό για τη στρατηγική του ΦΠΑ θα είναι ένα σημαντικό έγγραφο για να ορίσει τη στρατηγική κατεύθυνση του συστήματο ΦΠΑ στην Ευρώπη. Όμω, αυτό που δεν θέλω είναι να λάβουμε αποφάσει τώρα και να κινδυνεύσουμε να βρεθούμε εκτό του θέματο που θα θέσει η στρατηγική του ΦΠΑ. Η άποψή μου είναι ότι η πράξη για την ενιαία αγορά δεν θα πρέπει να κάνει συστάσεις για τους φόρους ή για αναθεωρήσεις ε, του συστήματος. Θα πρέπει να ενισχύσει τη στρατηγική του ΦΠΑ με κύριο σκοπό να καταπολεμηθεί η απάτη. Ευχαριστώ για τα σχόλια του κυρίου αυτό που έλεγα είναι ότι η πρόταση της Επιτροπής θα ήθελα να δημοσιευτεί πριν το 2013. Όχι πριν το 2013, μάλλον ως το 2013. Γι' αυτό μπόρεσα και να δεχτώ την τροπολογία του κ. Τάλερ. Γιατί έλεγα ότι ως το 2013 θα πρέπει να έχει γίνει η πρόταση της Επιτροπής. Όχι να ισχύει και η οδηγία. Και για, την τροπολογία, για τις τροπολογίες του κυρίου Τάλερ αυτό που μας λέει είναι ότι ή δυνατόν θα πρέπει να περάσουμε σε ένα οριστικό καθεστώς ως το 2015. Ή δυνατόν. Δεν νομίζω ότι καταναγκάζουμε κανέναν σε κάτι. Ούτε με την εκτροπολογία έχω ιδιαίτερη αντίρρηση. Απλώ να ευχαριστήσω του συναδέλφου για τη στήριξή του και ελπίζω ότι σύντομα θα γίνει η ψηφοφορία και ότι θα κλείσει και το θέμα ευνοϊκά. Να θυμίσω στου συναδέλφου ότι 9 Νοεμβρίου έχουμε την ψηφοφορία και στη δεύτερη ολομέλεια του Νοεμβρίου την ψηφοφορία. Την τελική. Ε, έχουμε προχωρήσει γρήγορα. Περνάμε λοιπόν στην έκθεση του κυρίου Ράπκαη για την ε, ονισμό του Συμβουλίου για τι κρατικέ ενισχύσει που διευκολύνουν την πάυση λειτουργία διαγωνιστικών ανθρακοριχείων. Κύριε Ράπκαϊ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε, ξέρετε όλοι εξάλλου συνάδελφοι ότι στις 27 ε, Σεπτεμβρίου ξεκίνησα την παρουσίαση του θέματος αυτού. Έλαβα κάποιες τροπολογίες για την πρόταση της Επιτροπής. Εν τω μεταξύ η προθεσμία έληξε για την ε, υποβολή των τροπολογιών. 72 τροπολογίες ε, έχω πάρει και τόσα χρόνια που βρίσκομαι εδώ στο Κοινοβούλιο, συνήθως όταν υπάρχουν τόσες πολλές ε, τροπολογίες, ε, θεωρούμε ότι το περιεχόμενο είναι ένα περιεχόμενο αμφισβητούμενο. Αν κοιτάξει κανείς ε, το θέμα αυτό και το περιεχόμενο, διαπιστώνουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι προφανές. Οι 70 από τις τροπολογίες στηρίζουν, αν θέλετε, την κατεύθυνση του κειμένου και μόνο δύο είναι καθαρά αμφισβητούμενες και αντίθετες. Θα ήθελα λοιπόν να πω ποια είναι η βάση του δικού μου σχεδίου έκθεσης. Όσον αφορά την αξιολόγηση αντικτύπου, Κάτι που πραγματικά με οδήγησε στην εξέταση του περιεχομένου της πρότασης της Επιτροπής. Διαπιστώνει κανείς ότι τα συμπεράσματα της Επιτροπής είναι, αν θέλετε, τελείως ε, διαφορετικά από αυτά στα οποία ε, κανονικά θα έπρεπε να φτάσουμε. Και αυτό, όπως ξέρετε, δεν είναι περίεργο, καθότι ο αρμόδιος ε, επίτροπος, ο κύριος Αλμούνια, για το θέμα των ε, επιδοτήσεων, προτείνει κάτι τελείως διαφορετικό από ότι το κολέγιο των επιτρόπων. Τους οι υπόλοιποι επίτροποι, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν διαφορετική κατεύθυνση. Ο, η εξέταση, λοιπόν, αντικτύπου φαίνεται να ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση η πρόταση της Επιτροπής που αναφέρει σαν ε, καταληκτική ημερομηνία το 2014 είναι κάτι το οποίο εδώ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμβαδίσει. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει το 2018 και σε αυτή την περίπτωση μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι δεν είναι συμβατά αυτά τα επιχειρήματα. Όταν υπάρχουν ε, βεβαίως τέτοιου είδους ε, συμμαχίες φτάνουμε σε τέτοια μη λογικά αποτελέσματα. Από τη μία λοιπόν υπάρχει ο κύριος Σαλμούνια και από την άλλη η ε, άποψη της Επιτροπής. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα ανταγωνισμού. Δεν πρόκειται για θέμα που αφορά την πολιτική περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντολογικές πτυχές βεβαίως πρέπει να ληφθούν υπόψη. Υπάρχει και η αντίστοιχη νομοθεσία. Εδώ όμως μιλάμε για ένα θέμα που αφορά περισσότερο τις ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις στον τομέα του άνθρακα και βεβαίως υπάρχουν και περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Αν θέλετε, η συνέπεια του περιορισμού χρήσης του άνθρακα σίγουρα ενδεχομένως είναι λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και την ίδια ώρα βλέπει κανείς ότι πρόκειται για μια πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη βιομηχανία, για τη χημεία. Ε, είναι λανθασμένο το συμπέρασμα και ένα δεύτερο λανθασμένο συμπέρασμα είναι η αντικατάσταση του άνθρακα στην Ευρώπη από άνθρακα ο οποίος εισάγεται. Και στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι σε ένα θέμα που αφορά τις επιδοτήσεις, τα στοιχεία αυτά δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Η αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν την μεγαλύτερη χρονική διάρκεια θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί γιατί και εδώ αυτά τα επιχειρήματα δεν συμβαδίζουν 100% με το θέμα των επιδοτήσεων. Τρίτη παρατήρηση που δεν θέλω να κάνω, θέμα ανταγωνισμού, θέμα επιδοτήσεων. Υπάρχει μία πρόταση η οποία λέει ότι δεν θέλουμε να υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Η Επιτροπή όμως, και αυτό το λέω για να σας το υποθυμίσω, ότι οι επιδοτήσεις για πάυση λειτουργίας για παραγωγή 2014, ο Επίτροπος Αλμούνη αναφέρεται στο 2018. Αντίθετα, ο κανονισμός αυτός έχει ισχύ ως το 2026, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι περιβαλλοντολογικές και οικονομικές συνέπειες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει και η πρόταση για καμία καταληκτική ημερομηνία, καμία προθεσμία. Βλέπουμε όμως ότι η νομολογία του δικαστηρίου μέχρι τώρα αναφέρει ότι θα πρέπει οι επιδοτήσεις να μειώνονται στο χρόνο και θα πρέπει να υπάρχει προθεσμία, καταληκτική ημερομηνία. Αυτή είναι η πάγια νομολογία του δικαστηρίου. Και πιστεύω ότι το 2026 είναι μια θεωρητική ημερομηνία, γιατί οι επιδοτήσεις έχουν έναν χαρακτήρα στήριξης από τις κρατικές αρχές προς τις επιχειρήσεις. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα θετικό κίνητρο, μια δυνατότητα στήριξης ή περιορισμού μιας πολιτικής. Και βεβαίως δεν δίνονται καμία, δεν δίνεται καμία επιδότηση, καμία στήριξη σε επιχειρήσεις αυτές οι οποίες πλήττουν το περιβάλλον ή έχουν αρνητικές κοινωνικές συνέπειες. Γι' αυτό και βεβαίως λαμβάνουμε υπόψη μας εδώ και την πολιτική στον τομέα της απασχόλησης. Μια τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω σήμερα το πρωί είναι αυτή που ανέφερε η πρόεδρος της ε, Νομικής Επιτροπής μαζί μου όταν μιλήσαμε για το θέμα της νομικής βάσης. Είναι το άρθρο 107. Εδώ όμως δεν περιέχεται η υποχρεωτική, η υποχρεωτική διαβούλευση. Αυτό ουσιαστικά το αποφάσισε το Συμβούλιο να υπάρξει διαβούλευση, αλλά αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική η διαβούλευση. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να επικαλεστούμε μάλλον το άρθρο 109. Όπως ξέρετε, η νομική βάση μπορεί να άλλαξε, γιατί ήταν η συνθήκη της Νίκιας, έχουμε περάσει στη Λισαβόνα Ίσως λοιπόν έχει αλλάξει και ο το άρθρο της νομικής βάσης. Θα πρέπει λοιπόν στην Λονομέλεια να είμαστε προσεκτικοί και προηγουμένως να ψηφίσουμε ποια θα είναι η νομική βάση. Και άλλη μία τελευταία ε, παρατήρηση, κύριε, κυρία Πρόεδρε. Μία παρατήρηση όσον αφορά την συνάντηση που έχουμε προβλέψει μεταξύ των ε, εισηγητών, σχεδόν εισηγητών και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μια ημερομηνία η οποία να μπορούν να δεχτούν όλοι. Εγώ ήρθα σε επαφή με όλους τους σχεδόν εισηγητές και πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να μπορέσουμε να βρούμε μια ημερομηνία στην οποία να συζητήσουμε όλες αυτές τις ε, προτάσεις. Πρέπει να συζητήσουμε και το κείμενο και βεβαίως το κείμενο αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι προβληματικό. Εγώ μπορώ να αποσύρω κάποιες από τις προτάσεις μου από τη στιγμή που τα άτομα αυτά που έχουν υποβάλει τροπολογίες θέλουν να γίνουν δεκτές οι τροπολογίες τους σε αντικατάσταση του κειμένου. Το συζήτησα αυτό με τους σκιώδες εισηγητές. Και πρέπει να σας πω ότι το συμπέρασμα στο οποίο φτάσαμε είναι ότι από τη στιγμή που δεν θέλουμε να αλλάξει το κείμενο. Και από τη στιγμή που πάνω από το 95% των τροπολογιών στηρίζουν ε, την ουσία του κειμένου, θα προτείνω εγώ ένα κείμενο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις τροπολογίες. Να μπορέσουμε να βρούμε δηλαδή μια συμβαστική λύση. Η συμβαστική αυτή λύση όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να λάβει υπόψη το 2014 ή 2013 και την καταληκτή ημερομηνία 2018. Μεταξύ αυτών βεβαίως των δύο προτάσεων δεν μπορεί να υπάρξει ε, συμφωνία. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ εγώ να βρω συμβιβαστική λύση μεταξύ του αν θα βρεθούν άνεργοι αυτοί οι άνθρωποι ή όχι. Μεταξύ των ανέργων και των μη ανέργων δεν υπάρχει συμβιβαστική λύση. Κατά τα άλλα, πραγματικά το κείμενο δεν είναι προβληματικό και πιστεύω ότι αν μπορούμε να αποφύγουμε την συνάντηση στην οποία δεν θα είναι όλοι οι εισηγητές, αυτοί που έχει προβληθεί για αύριο, ε, τόσο το καλύτερο, γιατί πραγματικά θα πρέπει να προχωρήσουμε με μια επικοδομητική διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ σαφής, ε, λέει η Πρόεδρος, η παρουσίασή σας καταλαβαίνουμε ποια είναι η θέση του εισηγητή, έχουμε και τους σκιώδες. Η... η κυρία Νέντβιλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί οι φιλελεύθεροι θα προτιμούσαν να υποστηρίξουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμφωνούμε με τις αλλαγές που προτείνει ο κύριος Ράπκαη και θα πρέπει να πω εδώ ότι εξορισμού δεν θα υποστηρίξουμε καμία από τις τροπολογίες γιατί πηγαίνουν ακόμα παραπέρα από αυτό που προτείνετε εσείς ως αλλαγή. και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγέ σε μία νυχτή. Δεν είναι πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο προέκυψε χθε. Είναι κάτι το οποίο συζητώνταν εδώ και χρόνια, μην σα πω και δεκαετίε. Και νομίζω ότι οι τομεί είχαν αρκετό χρόνο να κάνουν τι ανάλογε μεταρρυθμίσει και σε κάποιε χώρε έγιναν αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Επομένω, δεν είναι λογικό να. Ε, επιβραβεύσουμε κάποιες χώρες οι οποίες δεν έκαναν τις μεταρρυθμίσεις και να τιμωρήσουμε άλλες οι οποίες έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να γίνει. Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ προσεκτικά πού διαθέτουμε τα χρήματά μας και κατά πόσον θέλουμε να πληρώσουμε για τα προβλήματα του παρελθόντος ή να επενδύσουμε τα ευρώ μας στις προκλήσεις του μέλλοντος. Οι φιλελεύθεροι επιλέγουν τη δεύτερη επιλογή, κυρία Πρόεδρε. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι ούτως ή άλλως ε, θεωρούμε ότι πρόκειται για συμβιβασμό. Ε, θεωρούμε όμως ότι είναι ένας συμβιβασμός που μπορούμε να αποδεκτούμε, αλλά δεν θα θέλαμε να υποστηρίξουμε καμία επιπλέον αλλαγή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλούτερ από την... Ε, Ευχαριστώ. Εγώ θα πάρω διαφορετική θέση από την ε, συνάδελφο που μόλις μίλησε. Εγώ στηρίζω την πρόταση του κυρίου Ράπκαη. Η δική μας πρόταση ήταν 2020 προθεσμία, αλλά μπορώ να δεχτώ το 18, το 2018. Κατά τα άλλα δεν έχω άλλες παρατηρήσεις. Μπορώ να στηρίξω ε, την ε, πρόταση αυτή. Όσον αφορά την ημερομηνία 2018, η Γερμανία και η Ισπανία, όπως ξέρετε, πλήττονται άμεσα από το θέμα αυτό και βεβαίως πρέπει να ξέρετε ότι στην ε, Γερμανία οι πολιτικοί εκπρόσωποι και όλος ο τομέας ε, των ε, ανθρακοριχείων έχουν συνάψει μια συμφωνία από το 2006 για το 2018 και Αυτή η ημερομηνία το 2008 σαφώς και θα πρέπει να τηρήσει αυτήν την συμφωνία που έχει γίνει στη χώρα μας μεταξύ των ενδιαφερόμενων του τομέα αυτού. Δεν μπορούμε λοιπόν σε καμία περίπτωση να δεχτούμε κάτι ε, μία ημερομηνία πριν. Το θέμα του ανταγωνιστικού, αν θέλετε, επιχειρήματος. Δεν είναι δυνατόν εδώ να βασιστούμε μόνο στο θέμα της ανταγωνιστικότητας. Ο άνθρακας είναι μία πρώτη ύλη. Βεβαίως και θα πρέπει να αντικατασταθεί, μπορεί να αντικατασταθεί, αλλά για αυτό χρειάζεται μία πολιτική, αν θέλετε, διαδικασία, χρειάζεται συγκεκριμένη ασφάλεια και τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα αποθέματα του άνθρακα, γιατί δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι θα αντικατασταθεί ο άνθρακας χωρίς να έχουν βρεθεί προηγουμένως άλλες εναλλακτικές πηγές. Την ίδια ώρα έχουμε αυτά τα αποθέματα και η πρόσβαση σε αυτά τα αποθέματα θα πρέπει να παραμείνει ε, ελεύθερη και θα πρέπει πραγματικά επαναλαμβάνω να κοιτάξουμε το θέμα αυτό όχι μόνο από την άποψη του ανταγωνισμού αλλά από γενικότερη πολιτική άποψη και τεχνολογική. Ο κύριος Λάγκεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να πω ότι στηρίζουμε πλήρως την έκθεση του κυρίου Ράπκαη. Υπάρχουν κάποιες ε, διαφορετικές απόψεις σε κάποια σημεία, τις οποίες όμως ε, σε εσωτερικό επίπεδο θα συζητήσουμε και θα λύσουμε. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες όσον αφορά την ημερομηνία 2020, νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε το 2018. Εγώ τουλάχιστον θα στηρίξω την ε, ημερομηνία αυτή, την πρόταση αυτή στην πολιτική μας ομάδα. Τώρα, πρόκειται για θέμα ανταγωνισμού. Η Επιτροπή καλείται εδώ να αποφασίσει για ένα θέμα ανταγωνισμού. Εξού και ο Επίτροπος Αλμούνια πρότεινε το 2018 βασιζόμενος σε πολύ συγκεκριμένα επιστημονικά και τεκμηριωμένα στοιχεία. Η Επιτροπή γιατί δεν το δέχτηκε διότι υπήρξαν σκέψεις και θέματα που αφορούσαν πολύ περισσότερο το περιβάλλον, την, το κλίμα. Εδώ πρόκειται όμως καθαρά για θέμα ανταγωνισμού και πρόκειται για μία μεταβατική περίοδος η οποία βάσει της στήριξης από κρατικές, από εθνικές ε, πηγές θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα αυτά τα ανθρακοριχεία και όλο το κοινωνικό, αν θέλετε, αντίκτυπο. Εμείς εδώ, επαναλαμβάνω, είπαμε ότι το θέμα αυτό μας αφορά από άποψη ανταγωνισμού. είμαι 16 χρόνια εδώ και ασχολούμαι με το θέμα αυτό και ξέρετε πολύ καλά ότι ο το θέμα των αρμόδιων ταμείων είναι κάτι και ταμιευτηρίων συγγνώμη είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μην το δούμε με διαφορετικό τρόπο. Ο αρμόδιος επίτροπος για τον ανταγωνισμό εκφράστηκε εδώ πραγματικά γνωρίζοντας όλα αυτά τα θέματα. Και μην ξεχνάτε ότι όσον αφορά τις επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος, επί του κλίματος, δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Έχουμε εδώ μονάδες οι οποίες ε, τροφοδοτούνται είτε από τον άνθρακα τον ευρωπαϊκό ο οποίος προέρχεται από τα ευρωπαϊκά ανθρακοριχεία, είτε από άνθρακα ο οποίος εισάγεται από τον Καναδά ή από αλλού. Και μιλάω γιατί η χώρα μου έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Και κάνω μια έκκληση προς όλους τους συναδέλφους. Θα πρέπει πραγματικά να στηρίξουμε την πρόταση του κυρίου Ράπκαη και να δούμε το θέμα και από την άποψη της αλληλεγγύης και βεβαίως του ανταγωνισμού. Κυρία Γουίνπερ, έχω κάποια σχόλια από πλευρά του κυρίου Στρέτσεκ, ο οποίο ε, παρακολουθεί το θέμα εκ μέρου μα, αλλά δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Αλλά λίγο πολύ συμφωνούμε με τα όσα είπε και το ΕΛΚ και υποστηρίζει ο κύριο ε, Τράσεκ τα σχόλια του κυρίου Λάγκε. Επίση, τα σχόλια που ακούσαμε από του φιλελευθέρου σήμερα το πρωί είναι θέμα ανταγωνιστικότητα. Η ανταγωνιστικότητα είναι αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει και δεν θα πρέπει να το λησμονεί κανεί από εμά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σαφέ μήνυμα που προκύπτει. Όσο έχει η έκθεση θα μπορούσε να τη δεχτεί, αλλά θεωρεί ότι τα θέματα ανταγωνισμού θα πρέπει να επισημαίνονται και δεν θα πρέπει να λησμονούνται σε καμία περίπτωση. Η κυρία Μουνίθ Συγγνώμη, δεν είπα σωστά το όνομά σας. Ευχαριστώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα μιλήσω εξ ονόματος των Ισπανών Σοσιαλιστών. Ξέρετε ότι ο συνάδελφος, ο οποίος είναι μέλος εδώ στην Επιτροπή μας, ε, χρειάστηκε να φύγει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να γίνει υπουργό στην Ισπανία. Η αντιπροσωπεία των σοσιαλιστών της Ισπανίας υποστηρίζει απόλυτα την έκθεση ΡΑΠΚΑ ή θεωρούμε ότι είναι μια υπεύθυνη έκθεση οποία ανταποκρίνεται στην κρίσιμη κατάσταση του άνθρακα στην Ευρώπη διότι πρόκειται για τη μόνη ε, πηγή, αυτόχθονη πηγή ενέργειας για μας. Γι' αυτό λοιπόν έχετε την πλήρη υποστήριξη της Ισπανικής Αντιπροσωπείας ε, για την έκθεση ΡΑΠΚΑΙ. Παρουσιάσαμε παρόλα αυτά μια σειρά από τροπολογίες, ε, οι οποίες θεωρούμε ότι χρειάζονται για να επισημανθούν κάποια στοιχεία. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε λίγο περισσότερο τη σημασία των αυτόχθονων πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι σε κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μόνο άνθρακας ως ε, αυτόνομη πηγή και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ε, στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει σημείο κίνησης για να αναλύσουμε τις ε, κρατικές ενισχύσεις. Δεύτερον, όπως λέει και ο Μπέρναρ Ράπκα στην έκθεσή του, οι κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να παραμείνουν όχι μόνο για το κλείσιμο, για την πάυση λειτουργία, αλλά και για την μετάβαση σε έναν πιο ανταγωνιστικό τομέα που θα επιτρέψει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί εν γέννη. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει στις τροπολογίες να αναφέρεται ότι ρητά ότι θα πρέπει να υπάρχουν ενισχύσεις για έρευνα, για αλλαγή σε πιο καθαρές ε, ενέργειες και επίσης θα θέλαμε να προσθέσουμε στην έκθεση του Μπέρναρ Ράπκαϊ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνένεση εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, εμείς ε, θα μπορούσαμε να δεχτούμε να ε, παραταθεί η προθεσμία μέχρι το 2020 και να πρέπει να υπάρχει και κάποια σύνδεση ε, με κοινωνικού και περιβαλλοντικού παράγοντε. Να υπάρχουν δηλαδή κάποια ελάχιστα κριτήρια περιβάλλοντο και ε, κοινωνική ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Και επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ρητός και η ανάγκη να υπάρχει ένα στρατηγικό απόθεμα στην Ευρώπη, διότι ο άνθρακας, όπως είπα επανειλημμένως, είναι η μόνη αυτόνομη πηγή ενέργειας που έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη παραγωγή άνθρακα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προθεσμία πάυσης λειτουργίας, να υπάρχει μια μικρή πρόβλεψη για την περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα ενέργειας στην Ευρώπη. Αν κλείνει ένα ανθρακοριχείο και δεν υπάρχει δυνατότητα να ξανανοίξει, θα πρέπει να εξετάσουμε τουλάχιστον το ενδεχόμενο να μείνουν ανοιχτά κάποια ανθρακοριχεία για να υπάρχει τουλάχιστον ένα στρατηγικό απόθεμα ε, άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Okay, um, uh, ναι μου ζητήθηκε τελευταία στιγμή να προεδρεύσω συνεδρίες και δεν ήθελα να κάνω σχόλια ως πρόεδρος, θα κάνω σχόλια λοιπόν ως μέλος. Θα πω κάποια σχόλια τα οποία κατά πάσα πιθανότητα συμπίπτουν με κάποια από όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Πρέπει να υπάρχει υποστήριξη για θέσεις εργασίας και απασχόληση, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι η έβδομη παρέκκληση που δίνουμε στους ανθρακορίχους, είναι η έβδομη φορά που δίνεται αυτή η παρέκκληση και στα πλαίσια της πολιτικής ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα έννοιο καθεστώς ε, εξαιρέσεων. Καταλαβαίνω ότι είναι αυτά που λέτε κύριε Ράπκαη, αλλά εδώ υπάρχει πολιτική για τις ε, κλιματικές αλλαγές. Ε, κατανοώ ότι εσείς έχετε διαφορετική μέθοδο και διαφορετικά στοιχεία, Κύριε Λάγκεν, σας παρακαλώ μην διακόπτετε. Και επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια αξιόπιστη ημερομηνία. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού για τις προθεσμίες. Εγώ θα μπορούσα να δεχτώ μια νωρίτερη προθεσμία, εάν δεχτείτε να μην ε, διαγράψετε τις αναφορές ε, για το μετριασμό των αλλαγών του κλίματος. Και όπω είπε και η Ισπανίδα συνάδελφο, θα πρέπει να εξετάσουμε και κάποιε κρατικέ ενισχύσει για να κάνουμε μετατροπή σε πιο καθαρέ πηγέ ενέργεια. και αυτό φυσικά θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη για περιβαλλοντικού λόγου. και αν εστιάζουμε απλώ και μόνο στο θέμα τη πολιτική ανταγωνισμού, είναι πολύ σημαντικό η ενίσχυση που δίνεται για την υποστήριξη των ανθρακοριχείων στο μέλλον να μην ε, είναι εις βάρος ε, του ανταγωνισμού για χώρες οι οποίες δεν βασίζονται και δεν στα ανθρακοριχεία και δεν έχουν αθέμητο ανταγωνισμό σε φτηνή παραγωγή ενέργειας. Όπως και να το εξετάσουμε, εξακολουθεί να είναι ένα θέμα ε, ουσιαστικά ανταγωνισμού, το οποίο φυσικά έχει και κάποιες άλλες πτυχές. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε έναν ε, λογικό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Δεν θέλουμε να έχουμε ανέργους, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε τις, εξετάσεις, τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τρόπον ώστε να έχουμε μια λογική πρόταση για την πάυση λειτουργίας των ανθρακοριχείων, αλλά εάν δεν κλείσουν και είναι κερδοφόρα θα πρέπει ε, να επιστρέφουν την κρατική ενέργη, ενίσχυση ε, στα πλαίσια της πολιτικής ανταγωνισμού. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε το θέμα. Ε, ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σεβασμό και ε, ο εισηγητή και οι σκιώδει εισηγητέ να μην διαγράψουν όλε τι αναφορέ που έχουμε στι περιβαλλοντικέ αλλαγέ και στην ε, καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο. Μπορεί να χρειαστεί να παραταθεί το, η προθεσμία για την πάυση λειτουργίας, αλλά θα πρέπει τελικώς να υπάρξει μία πάυση. Τώρα αναλαμβάνω πάλι καθήκοντα Προέδρου και δίνω τον λόγο στον εισηγητή. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ε, απευθύνω λοιπόν το λόγο σαν μέλος της Επιτροπής και όχι σαν Πρόεδρος. Το θέμα βεβαίως είναι πώς ερμηνεύουμε τα στοιχεία. Αναφερόμαστε σε στοιχεία και θα ήθελα να πω με πολύ σαφή τρόπο. Αυτό που λέτε είναι ότι βεβαίως υπάρχουν επιπτώσεις στο κλίμα, στο περιβάλλον. Μα εννοείται, το κάθε θέμα που αφορά την ενέργεια έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, στο κλίμα. Και το θέμα είναι ότι εάν πάρουμε μέτρα που αφορούν την παραγωγή άνθρακα στην Ισπανία, στη Γερμανία, στην Ρουμανία και στην Ουγγαρία, γιατί αυτές είναι οι χώρες τις οποίες πλήττει αυτό το κείμενο, ουσιαστικά θα έχει το εξής αποτέλεσμα. Κάθε σταμάτημα της παραγωγής από ανθρακοριχία της Ευρώπης, αυτών των τεσσάρων χωρών, θα αντικατασταθεί από άνθρακα που εισάγουμε από μία τρίτη χώρα. Το ε, αποτέλεσμα λοιπόν επί του περιβάλλοντος θα είναι μηδανικό. Αυτό είναι. Πρόκειται λοιπόν καθαρά για θέμα ευρωπαϊκής πολιτικής, ασφάλειας, πρόκειται για μια πηγή ενέργειας και θα ήθελα να πω στην συνάδελφο Ινφελτ περιγράφουμε τον άνθρακα σαν ένα προϊόν του παρελθόντος. Αυτό όμως δεν ισχύει πια. Και σήμερα βλέπουμε ότι ο άνθρακας παγκοσμίως αντιμετωπίζεται με τελείως διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση του άνθρακα σε σχέση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και η σημασία του άνθρακα αυξάνεται, διαφοροποιείται ο άνθρακας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και βεβαίως είναι θέμα τεχνολογίας από εκεί και πέρα. Πώς θα δημιουργήσουμε ηλεκτρική ενέργεια με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν τεχνολογίες που μας οδηγούν στην καθαρή καύση του άνθρακα. Αυτές θα πρέπει να αναπτύξουμε και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε το κλίμα και το περιβάλλον και εκεί. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι όταν λέτε ότι υπάρχουν χώρες που δεν έκαναν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Κοιτάξτε αγαπητοί συνάδελφοι. Πρόκειται για χώρες που βεβαίως ξεκινάνε από τελείως διαφορετικά επίπεδα. Μιλάμε για χώρες που είχαν 200.000 θέσεις απασχόλησης και έφτασαν στο μηδέν. Άλλες χώρες ξεκινάνε από 600.000. Είναι λοιπόν θέμα επίπεδου εκκίνησης. Είναι θέμα εύκολων ή πολύ πιο δύσκολων αναδιαρθρώσεων και κοινωνικών συνεπειών πολύ πιο σημαντικών. Και υπάρχουν θέματα που αφορούν πολύ περισσότερο κάποιες χώρες και τα μέτρα αυτά τα συνοδευτικά, όπως καταλαβαίνετε, που αφορούν τον τομέα των ε, ανθρακοριχείων ε, στην Γερμανία, αφορούν και την Ισπανία. Εγώ θα επισκεφτώ την Ισπανία και θέλω να δω πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Αύριο θα συναντηθώ και με εκπροσώπους του τομέα από την Ισπανία. Το λέω αυτό γιατί δεν έχω αυτή την ευαισθησία και δεν ασχολούμαι με το θέμα αυτό μόνο επειδή είμαι Γερμανός. Πιστεύω πραγματικά ότι ακριβώς αυτό που πρότεινε ο αρμόδιος επίτροπος για τον ανταγωνισμό είναι κάτι που θα πρέπει να μας ε, οδηγήσει στην κατεύθυνση και στον προσανατολισμό αυτό στον οποίο όλοι συμφωνήσαμε. Οι ενισχύσεις θα πρέπει να είναι ενισχύσεις που μειώνονται στο χρόνο. Θα πρέπει να έχουν μια καταληκτική ημερομηνία και πραγματικά θέλω να σας πω ότι εγώ παρακολουθώ το θέμα αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη ήμουν εισηγητής το 2002. Ξέρω ποια είναι τα επιχειρήματα όλων και ποια είναι το ενδιαφέρον όλων και η καταληκτική ημερομηνία, όπως σας είπα, θα πρέπει να βασιστεί στην πάγια νομολογία και στις αποφάσεις του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου. Οι ενισχύσεις θα πρέπει να περιορίζονται και θα πρέπει να υπάρχει και μια καταληκτική ημερομηνία. Και θα πρέπει να έχουμε ένα σημείο στον ορίζοντα, τον οποίο να προσβλέπουμε και όπως ξέρετε και σε άλλους τομείς υπήρξαν ε, ενισχύσεις οι οποίες ε, τελικά επιμικύνθηκαν στο χρόνο. Η διαφορά όμως μεταξύ αυτού και του νέου κανονισμού είναι ότι ο κανονισμός ο οποίος λύγει σε καμία περίπτωση δεν αναφέρει τη σημερινή κατάσταση σε σχέση με την καταληκτική ημερομηνία. Εδώ αναφερθήκαμε στο 2018. Το 2018 είναι κάτι που δεν το αμφισβητούμε με την έννοια ότι αναφέρατε και εσείς ε, κυρία Πρόεδρε το θέμα των ανταγωνιστικών ανθρακοριχείων. Τι θα γίνει με τις περιπτώσεις αυτές όπου η παραγωγή άνθρακα είναι ανταγωνιστική. Γιατί σε μια κανονική διαδικασία ενισχύσεων η επιχείρηση η οποία δεν ήταν ανταγωνιστική, σώθηκε όμως, ενισχύθηκε και έγινε ανταγωνιστική, πρέπει να επιστρέψει όλα τα ποσά που είχε λάβει. Γιατί λοιπόν εδώ προτείνουμε κάτι τέτοιο. Αυτά. Κατά τα άλλα, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να συζητήσουμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία με την κυρία Ίνφελ. Για κάποια άλλα δεν υπάρχει συμβιβασμός. Επαναλαμβάνω ότι οτιδήποτε ημερομηνία πριν το 2018 σημαίνει για τη γερμανική, την ισπανική και άλλες βιομηχανίες, για άλλους χώρες μεγάλο αριθμό ανέργων. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Και όπως είπα και στην αρχή της παρουσίασής μου θα προσπαθήσω να συναντήσω τους σκιώδεις εισηγητές και πιστεύω ότι πολύ σύντομα για τα άλλα σημεία θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Κυρία Ινφελτ, πολύ σύντομα πρόεδρε, μπορεί να διαφωνούμε για τα πολιτικά ζητήματα, όμως δεν μπορώ να δεχτώ την ε, πρόταση ότι δική μας η θέση αυτομάτως οδηγεί σε απολύσεις εσείς πολύ σωστά ως μέρος της Επιτροπής ε, ε, επισημάνατε ότι είναι η έβδομη απόφαση να παραταθούν από οι νέες διαθετήσεις. Δεν είναι ένα πρόβλημα που προέκυψε χθε. Δεν μπορείτε να λέτε ότι επειδή διαφωνούμε με την ε, περαιτέρω παράταση οποιαδήποτε απόλυση θα ήταν δική μας ευθύνη. Όχι, με συγχωρείτε. Εάν πρέπει να αποφασίσουμε κάτι ανάλογο για τον τομέα των τραπεζών, να επιδοτήσουμε τον τραπεζικό τομέα για δεκαετίες επί δεκαετιών εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Εάν μιλάμε λοιπόν για μια βιομηχανία για το μέλλον, δεν θα έπρεπε να χρειάζεται τόσες επιδοτήσεις για τόσες δεκαετίες στην Ευρώπη. Μάλιστα, ήταν έντονη η συζήτηση. Νομίζω ότι όλο αυτό εντάσσεται και στο θέμα τη φορολόγηση του χρηματοστατικού τομέα. Κύριε Λάγκε, θέλετε επανέλθετε πολύ σύντομα. Μια σύντομη παρατήρηση. Οι ενισχύσει για τον τομέα του άνθρωκα είναι χαμηλότερη σε σχέση με την διάσωση μιας ε, Ολλανδικής τράπεζας. Ε, κοιτάξτε τα ποσά και συγκρίνετε τα. Ναι, όπως λέτε, οι επιδοτήσεις για τον τραπεζικό τομέα έχουν φτάσει στα δισεκατομμύρια κάποιες περιπτώσεις, αλλά κάποια στιγμή ελπίζουμε θα τα πάρουμε και πίσω. Τέλος πάντων, ενδιαφέρουσα η συζήτηση, θα ψηφίσουμε στις 9 Νοεμβρίου και θα πάμε στην ε, δεύτερη ολομέλεια του Νοεμβρίου. Νομίζω η συγκεκριτής μας απάντησε σε πολλά από τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσει να με συμβιβαστικέ λύσει, όπω είπαμε, και να δούμε κατά πόσο θα υπάρξει στήριξη για την πρότασή του. προχωρούμε λοιπόν τώρα στην έκθεση του κυρίου Στολόγεν. Τροπολογίε στι οδηγίε 98-78, δεν θα τι διαβάσω όλε. Συμπληρωματική εποπτεία λοιπόν των χρηματοπιστωτικών εντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων. Κύριε Στολόγεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε μπροστά μας μια πρόταση για μια οδηγία που αναθεωρεί τρεις οδηγίες για τη συμπληρωματική εποπτεία. Οι βασικές, η βασική οδηγία είναι η 2002 του η οποία επικεντρώνεται στη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ομήλων και έχουμε δύο ακόμη οδηγίες. Η μία για τη συμπληρωματική εποπτεία των ασφαλιστικών οντοτήτων μέλος ασφαλιστικών, μέρος ασφαλιστικών ομίλων και την οδηγία του 2006-48 για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στην πραγματικότητα ομιλούμε για χρηματοπιστωτικούς ομίλους με τέτοια πρότυπα που συνδυάζουν υπηρεσίες και προϊόντα επιχειρηματικά ε, σε διάφορες ε, φάσεις της ε, χρηματοπιστωτικής αγοράς. Δηλαδή τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, και ούτω καθεξής. Ο στόχος της οδηγίας αυτής, αυτής που πρόκειται να θεωρηθεί δηλαδή με την τωρινή πρόταση οδηγίας, είναι να ελέγξει τον ενδεχόμενο κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από την πολλαπλή χρήση των κεφαλαίων σε τέτοιες περιπτώσεις ομίλων και τον παρελκόμενο κίνδυνο που παρουσιάζει ο πολύπλοκος χαρακτήρας των ομίλων αυτών, η διαχείρισή τους, η συγκέντρωση, η σύγκρουση συμφορώντων και όταν η οδηγία του 2002-87, η βασική όπως είπα οδηγία, που εισάγει στο επίπεδο ομίλου την συμπληρωματική εποπτεία. Όταν εγκρίθηκε λοιπόν η οδηγία αυτή, η πρόθεση ήταν να υπάρξει θεώρηση μετά από κάποια χρόνια και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκόπευε να κάνει την αναθεώρηση σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι η τωρινή μας πρόταση οδηγία, η οποία επικεντρώνεται στα κατεξοχήν τεχνικά ζητήματα. Προέκυψε μάλιστα από, μια, από, από διάφορους γύρους διαβουλεύσεων, με υπευθύνωση των ασφαλιστικών εταιριών, του τραπεζικού τομέα, ε, λήφθησαν υπόψη αποτελέσματα Κροάσιων και ούτω καθεξής. Και έπειτα θα υπάρξει μια δεύτερη φάση που θα αναπτυχθεί μετά το 2010, ίσως του χρόνου, η οποία πρόκειται να περάσει σε μια πιο ριζική αναθεώρηση σε σχέση με το πεδίο, τα κεφάλαια και ούτω καθεξής. Οι πιο σημαντικές αλλαγές που επιφέρει αυτή η πρόταση οδηγίας είναι η εξή. Πρώτον, προσπαθεί να αποφύγει, να καλύψει κάποιες μαύρες τρύπες που υπήρχαν προηγουμένως από τις προηγούμενες οδηγίες και το βασικό ζήτημα ήταν ότι υπάρχουν διατάξεις και αρμοδιότητες για τις εποπτικές αρχές που μπορούν να ισχύσουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους, αλλά μόνον τομεακά. Όταν οι τραπεζικές δραστηριότητες ή ένας ασφαλιστικός όμιλος αλλάζει κατηγορία λόγω μιας εξαγοράς, μιας άλλης εταιρείας λόγω χάρη, από άλλον τομέα, και περνάει στην κατηγορία του χρηματοπιστικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, τότε οι, σημεριν, οι προηγούμενες οδηγίες αφήνουν κάποιες γκρίζες ζώνες, κάποιες αμφιβολίες για το τι γίνεται ακριβώς με την εποπτεία. Πώς η εποπτεία δηλαδή θα ισχύει για την ε, νέα εταιρεία, για το νέο όμιλο. Ε, δηλαδή υπάρχει ένα θέμα με την εποπτεία του τραπεζικού και του ασφαλιστικού σχέλους. Υπάρχει θέμα λοιπόν καλύτερου συντονισμού των ανάλογων ε, αρμόδιων αρχών που θα πρέπει να κάνουν την εποπτεία. Σε χώρες όπου υπάρχουν τραπεζικές αρχές, μάλλον υπάρχουν οι αρχές των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών, των υπουργείων, τα πάντα εξαρτώνται από το ποια χώρα, από ποια χώρα στη Σκοπιά βλέπουμε το θέμα. Ο στόχος λοιπόν είναι να υπάρξει καλύτερος συντονισμός όταν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος θα παρακολουθήσει, θα ελέγξει αυτούς τους σηματοποιητικούς ομίλους με τόσο πολλαπλές δραστηριότητες των, ε, στις επενδύσεις, στις, στα τραπεζικά, στα ασφαλιστικά. Η δεύτερη σοβαρή αλλαγή αφορά τον ε, εντοπισμό των χρηματοπιστωτικών ομίλων. Εδώ η σημαντικότερη πρόβλεψη είναι να συμπεριλάβουμε σε κάθε περίπτωση τις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η ισχύουσα οδηγία αφήνει μια τέτοια δυνατότητα, δεν ισχύει όμως υποχρεωτικά και δεν είναι σαφές ποια είναι τα κριτήρια που επιτρέπουν να αποφασιστεί ο χρηματοπιστωτικό όμιλο ποιο είναι. Επίση, υπάρχει ένα θέμα με τι κατευθυντηρίε γραμμέ που θα πρέπει να ισχύουν για τις εξαιρέσεις, εξαιρέσεις για μεγάλους ομίλους, ώστε να μην συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα της συμπληρωματικής εποπτείας. Στόχος εδώ είναι να επιτρέψουμε τον εντοπισμό μεν των χρηματοπιστωτικών ομίλων, αλλά να αποφύγουμε και καταστάσει όπου λόγω χάρη οι μικρότεροι όμιλοι θα πάγονται σε συμπληρωματική εποπτεία, ενώ οι γιγάντιοι κάποιες φορές όμιλοι θα εποφελούνται από την εξαίρεση. Υπάρχουν και άλλες αλλαγές που προτείνονται, όπως η επικαιροποίηση των ορισμών, η βελτίωση ή καλύτερα απλούστευση της μεθοδολογίας υπολογισμού του κεφαλαίου σε επίπεδο ομίλου και επίσης καθώς ήδη έχουμε νέες ευρωπαϊκές αρχές αρμόδιες όπως την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, την Ευρωπαϊκή Αρχή για τα ασφαλιστικά ζητήματα και τις συντάξεις και τις ισχύουσες οδηγίες για την εποπτεία και τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ομίλων, είναι απαραίτητο να παραπέμπουμε και σε αυτές τις νέες ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι αυτές οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν ακριβώς κατευθυντήρες γραμμές σε σχέση με την εποπτεία. Τα ζητήματα που εγώ ε, επεσήμανα σε σχέση με την πρόταση αυτή είναι τα εξή. Έχουμε, όπως ξέρετε, την οδηγία Solvency 2 που αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση και τα σχετικά ζητήματα και η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί από τα κράτη-μέλη από το 2012 φαίνεται ότι στη δική μας πρόταση οδηγίας υπάρχει παραπομπή στην οδηγία ε, Solvency 2. Η παραπομπή λοιπόν θα πρέπει να προσαρμοστεί στις αλλαγές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε σχέση με τις τωρινές οδηγίες. Επίσης για τη διαμεσολάβηση και τη διατησία και την συμπερίληψη ή όχι των οντοτήτων ε, στην ε, συμπληρωματική εποπτεία. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι κάποιος, μια αρχή ας πούμε, μπορεί να αποφασίσει αν θα συμπεριλάβει ή όχι έναν ε, όμιλο. Ίσως επίσης η διαιτησία είναι σημαντική για τις δραστηριότητες συντονισμού μεταξύ των διαφόρων αρχών που είναι υπεύθυνε για την εποπτεία. Οι ειδήσει τώρα που έχω από διαφορετικές συναντήσεις στο επίπεδο του Συμβουλίου, διότι το Συμβούλιο ήδη έχει καταπιαστεί με το θέμα αυτό σε κάποιες συναντήσεις και σε σχέση με αυτή την πρόταση οδηγία, φαίνεται να μην υπάρχουν σοβαρές ε, αντιπαραθέσει, σοβαρέ διαφωνίε στο επίπεδο του Συμβουλίου Α, ωστόσο ενημερώθηκα μετά από συζητήσεις με προσώπους κατών μελών ότι είναι αρκετά τα κρατημέλη που ζήτησαν από το Συμβούλιο να παρατείνει τις διορίες για την υλοποίηση σε επίπεδο κρατών μελών. Το Νοέμβριο θα συνεχίσω τη συνεργασία μου και τις συζητήσει με τους κοιότητες εισηγητές προκειμένου να ετοιμαστεί η έκθεση. Ίσως ε, ως το τέλος Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε κύριε Στόλογιαν ο κύριο Σκίνερ, εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον κύριο Στόλογιαν για τι παρατηρήσει του. Ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική η παρέμβασή σας ε, σε εν είδη του έργου που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει πραγματικά να δοθεί έμφαση σε αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση. Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείε που δρούν σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ως ασφαλιστικές εταιρείε αλλά και ως χρηματοπιστωτικοί όμιλοι. Αυτό λοιπόν κάποτε έχει αποσχολήσει ε, πολλούς συναδέλφου για το πώ οι εταιρείε κεφαλαίων μπορεί να ξεφύγουν από την εποπτεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που είναι πλέον πολύ επίκαιρο και απασχολεί ιδιαίτερα στο κοινό. Θα πληρώσουμε σοβαρό τίμημα εάν σύντομα δεν προσαρμοστούμε και δεν μπορέσουμε να εποπτεύουμε αυτού του μεγάλου ομιλού όπου υπάρχουν για την διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. όπω είπατε την τράπεζα, τα ασφαλιστικά για την πρόταση που έχει υποβάλει η Επιτροπή και προκειμένου να καλυφθούν μαύρε τρύπε μέχρι με την ε, προηγούμενη νομοθεσία. Ε, τις προάλλες ε, φαίνεται να συζητούσαμε κάτι ανάλογο και να είχαμε κάνει τις σχετικές προσαρμογές. Τώρα τα πράγματα πάλι έχουν, μας έχουν ξεπεράσει. Αλλά το θέμα είναι να αποτεμήσουμε το γενικότερο σκηνικό. Δηλαδή, όπως σωστά λέτε, η πιο συνετή στάση εδώ είναι να σκεφτούμε τις επιπτώσεις, διότι πολλές από τις συνεργασίες, πολλές από τις από τους συνδυασμού στον τομέα των χρηματοπιστωτικών ε, υπηρεσιών είναι ε, ιδιαίτερα περίπλοκη. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δράση γέρος και να είμαστε και αποτελεσματικοί. Ο ρόλος που θα μπορούσαμε να διαδραματίσουμε εμείς ως Κοινοβούλιο είναι να σκεφτούμε τι τροπολογίες μπορεί να επιφέρουμε ε, και να τις εξετάζουμε όσο προκύπτουν και εάν δούμε ότι δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, σοβαροί κίνδυνοι για την όλη κατεύθυνση της πρότασης, μπορούμε να συμπορευτούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικώ. Μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας ως προς το ότι οι διαπραγματεύσεις ως τώρα εδώ έχουν ε, φανεί αποτελεσματικές ε, για το, τη δέσμη της εποπτείας της χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και με την ΕΟΠΑ θυμάμαι πολύ καλά ότι είδαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίζουμε το τι αποφασίζουμε εμείς αμέσως ε, και το τι μέσους μπορεί να προκαλέσουν οι ε, αποφάσεις μας ως συνέπεια συνάδελφοι θα θυμούνται εδώ τις συζητήσεις που είχαμε για τη δέσμη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το τι νομοθετικές επιπτώσεις θα υπάρξουν από όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν εδώ δικό ρόλο να διαδραματίσουμε και πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτό το ρόλο μας μέσω της έκθεσης αυτής. Είναι πολλά αυτά που είναι κοινά στον τομέα των τραπεζών, των ασφαλίσεων, των κεφαλαίων. Θα πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσουμε τα διαφορετικά προϊόντα. Ε, και να ξέρουμε ότι αν θέλουμε να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη θα πρέπει να, αναλα... να ορίσουμε και τον κατάλληλο αρμόδιο για κάθε περίπτωση ώστε τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν υγιείς και εύρωστους τους ανάλογους τομείς. Στο επίπεδο λοιπόν των τριών επιτροπών, καθώ και σε συνεργασία με τι ευρωπαϊκέ αρχέ και του οργανισμού που πρόκειται να αρχίσουν να λειτουργούν, θα πρέπει να εμπλέξουμε στην όλη διαδικασία όλου αυτού του φορεί, καθώ και την ε, μεικτή επιτροπή, και να εκμεταλλευτούμε όλε τι ε, νέε ιδέε που προκύπτουν για το πώ θα ενισχύσουμε το ρόλο μα. Αυτό θα είναι το ζήτημα που θα πρέπει να μα απασχολεί. Τώρα, οι που με ανησυχούν κάπω είναι ότι η ίδια δέσμευση δεν φαίνεται να υπάρχει από του ε, υπευθύνου του μεγάλου αρχιτεκτονήματος των νέων αυτών ευρωπαϊκών αρχών. Εμείς τώρα ως βουλευτές θα πρέπει να τους ε, δεσμεύσουμε, να τους ε, προκαλέσουμε να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα ώστε να ασχοληθούν με καινοτόμε και επικοδομητικές ιδέες που θα επιτρέψουν σε αυτή τη βιομηχανία να προχωρήσει. Ελπίζω λοιπόν ότι θα συνεργαστούμε αποτελεσματικά και με του υπόλοιπου σκιώδε ώστε η υπόσχεσή μα και η αφοσίωσή μα να δώσουν τα κατάλληλα αποτελέσματα σε αυτή τη συγκεκριμένη νομοθετική πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίκολα από τις Παρασίνους. Ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι μετά από 8 χρόνια προσπαθούμε να κλείσουμε τα κενά. Είναι απαραίτητο πράγματι αυτό και συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια σειρά από σημαντικές από ε, παρατηρήσεις, τις οποίες θα πρέπει να συμμεριστούμε και εμείς. Θα ήθελα να θίξω βέβαια κάποια σημεία εδώ. Καταρχάς, υπάρχουν κάποια σημεία Ε, Παραδείγματο χάρη αναφέρεται η ΙΜΠΑ και η ΟΜΠΑ αλλά δεν αναφέρεται η ΕΣΜΑ. Καλό θα ήταν λοιπόν να αναφέρονται και οι τρεις αρχές αλλά και όχι μόνο οι δύο. Επίσης, συμφωνώ απολύτως με τον Πίτερ Σκίνερ για την κοινή επιτροπή. Θα πρέπει να είναι μια ισχυρή κοινή επιτροπή και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να την κάνουμε ισχυρή στα πλαίσια της οδηγίας αυτής. Η συζήτηση αυτή έχει γίνει και στο παρελθόν και κατ' εμέ δεν ολοκληρώθηκε και ποτέ. Ε, τώρα φτάνουμε στην τομεακή νομοθεσία και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή μας ε, θα διαδραματίσει ισχυρό αν όχι και ηγετικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο και θα πρέπει να ξαναρχίσει η συζήτηση. Διότι δεν είναι λογικό αυτό που έχουμε στην ε, ε, έκθεση ως θέση κάποιων κρατών μελών. Τρίτον, με ενδιαφέρει ο ρόλος των ε, οχημάτων ειδικών ε, σκοπών και αυτό θα πρέπει να το δούμε στα πλαίσια των ομίλων και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα συμπεριλάβουμε στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά σημεία τα οποία μας ενδιαφέρουν και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας ε, με το πνεύμα συνεργασίας που διέπει την όλη επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια η κυρία Σουίμπερν. Θα είμαι λακωνική. Συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα είπαν οι προλαλήσαντε. Ε, νομίζω ότι η αρχική εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλή και αποτελεί μια πολύ ισχυρή βάση εργασίας. Νομίζω ότι εκφύσεως ε, η οδηγία για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ε, και οι επιχειρήσεις που τη χρησιμοποιούν είναι το πρώτο τεστ, η πρώτη δοκιμή και θα πρέπει από εκεί και πέρα να δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Αν ενισχύσουμε λοιπόν τα όσα αφορούν στην κοινή επιτροπή, όπως έχω πει και στο παρελθόν, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δουλειά μας. Έχετε την πλήρη υποστήριξή μου λοιπόν για την κοινή επιτροπή ε, και θα πρέπει να δούμε πώς βλέπει το Κοινοβούλιο την αγαστή λειτουργία αυτών των τριών αρχών. Αν δεν συνεργαστούν θα έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα με αυτά τα ε, συστηματικά επικίνδυνα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την κοινή επιτροπή για να πληρώσουμε τα χάσματα τα οποία μπορεί να προκύψουν. Συμφωνώ λοιπόν και με τα σχόλια του Πίτερ Σκίνερ αλλά και με ε, του προηγούμενου συναδέλφου. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε και την ΕΣΜΑ. Είναι τρεις εποπτικές αρχές, έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες και αφορούν διαφορετικά προϊόντα. Επομένως θα πρέπει να λειτουργούν συλλογικά και οι τρεις αυτές επιτροπές και πολύ καλά στην Κοινή Επιτροπή όπως ακριβώς είχε προβληθεί όταν συστήθηκε. Θα σταματήσω εδώ γιατί νομίζω ότι υπάρχει γενικότερα συνένεση για το που θέλουμε να καταλήξουμε. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή για να ολοκληρώσει και να απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές και τους συναδέλφους um, που πήραν το λόγο συμφωνώ με το όλο σκεπτικό της ενίσχυσης του ρόλου της κοινή Επιτροπής και με κάποιες άλλες προτάσεις ε, που παρουσιάστηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης προς εξέταση στην ε, συνεδρίαση του Ιανουαρίου. Ε, οι προθεσμίες είναι κάπου στο Φεβρουάριο, να ψηφίσουμε δηλαδή ε, στην Επιτροπή 21 ε, Μαρτίου και μετά στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει αρκετός χρόνο στη διάθεσή μας για να το εξετάσουμε και να εξετάσουμε και κάποια από τα θέματα που παρουσίασε και ο εισηγητής και η Σκιώδης. Προχωρούμε. Είναι λίγο νωρίς, δεν ξέρω αν έχουν έρθει όλοι όσοι πρέπει να είναι εδώ. Είμαστε 10 λεπτά πριν από το κανονική ροή των εργασιών μας. Και τώρα έχουμε ένα σημαντικό πακέτο, μια δέσμη με 6 εισηγητέ, 14 σκιώδεις εισηγητέ και θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε επικοδομητικά το χρόνο μα. Ε, με ανησυχεί λοιπόν το γεγονό ότι δεν έχουμε εισηγητέ. Um, Να ζητήσω από τι πολιτικέ ομάδε να τηλεφωνήσουν στα γραφεία των εισηγητών για να του ζητήσουν να έρθουν και να προχωρήσουμε και εμεί με τι εργασίε μα στη συνέχεια.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 Θα συνεχίσουμε στις 11 γιατί δεν είναι εδώ οι συγητές. Ούτω Ούτως ή άλλως το πρόγραμμα ήταν για τις 11. Επομένως ε, θα κάνουμε ένα-δυο λεπτά διάλειμμα. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ έχει έρθει. Επομένως ο κύριος Φέιο, η κυρία Φερέιρα είναι εδώ, αλλά δεν έχουμε σκιώδεις συγητές. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ένα-δυο σκιώδεις, αλλά όχι όλους. Καθίστε συνάδελφοι να ξεκινήσουμε τώρα γιατί έχουμε μόνο μια μισή ώρα στη διάθεσή μας για να ασχοληθούμε με αυτό το περίπλοκο και πλήρες πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση. Όπως έλεγα πριν έρθουν και όλοι οι συνάδελφοι έχουμε έξι εισηγητές, 14 όδες εισηγητές και φαντάζομαι ότι και άλλοι θα ενδιαφέρονται να παρέμβουν και να ακούσουμε την άποψή τους για τη συζήτηση. Θα δώσω πέντε λεπτά στον κάθε συγητή. Θα σας χρονομετρώ για να υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχουν όλοι στη συζήτηση. Κατόπιν θα δώσω το λόγο στους κοιόδης συζητητές για τρία λεπτά περίπου ο καθένας και μετά και πάλι στους συζητητές και ε, θα τους δώσουμε άλλα δυόμιση λεπτά για να ολοκληρώσουν και φυσικά θα δώσω το λόγο και σε όλους όσους θέλουν να παρέμβουν στη συζήτηση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Καταρχάς να δώσουμε το λόγο στην κυρία Βόρτμαν Κόλ για την ε, ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Κυρία Βόρτμαν Κόλ, έχετε το λόγο. Yes, ε, thank you. Ναι, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Εμείς ως Κοινοβούλιο βρισκόμαστε στην έναρξη μιας ε, νομοθετικής ε, διαδικασίας ε, για έξι θέματα για την οικονομική διακυβέρνηση. Βέβαια για το Κοινοβούλιο δεν είναι η αρχή αυτή, διότι έχει γίνει αρκετή δουλειά, κυρίως στην έκθεση του Διόγκο Φέιο και στα πλαίσια της έκθεσης της κυρίας Μπερές. Επομένως, δεν ξεκινούμε από το μηδέν. Υπάρχει μια κοινή γραμμή από την οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε και να οικοδομήσουμε τη θέση μας. Είναι βέβαια λίγο περίεργη διαδικασία, διότι αν διαβάσει κάποιους εφημερίδες ε, και δει ε, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα ειδικών καθηκόντων, ε, δίνει την εντύπωση ότι την επόμενη εβδομάδα θα φτάσουμε στο τελικό σημείο, έχει τελειώσει, λες και έχει τελειώσει η συζήτηση και είμαστε όλα έτοιμα. Είναι καλό λοιπόν που οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων έδωσαν κάποιε σαφεί δηλώσει επί του θέματο αυτό την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, διότι μέχρι τούδα δεν έχει ληφθεί υπόψη η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή. Και ευτυχώ, μετά από την έναρξη λειτουργία τη συνθήκη Λισαβόνα, οι δέσμοι αυτοί των προτάσεων ε, είναι στη διαδικασία συνομοθέτη και επομένως μπορούμε να ακολουθήσουμε τη συζήτηση και βάσει των συζητήσεων που θα κάνουμε ε, με όλους τους συναδόλφους μπορούμε να εκπονήσουμε τις θέσεις μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό εφαλτήριο. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι να φροντίσουμε να έχουμε μια ταχεία διαδικασία, τουλάχιστον για την αρχή, διότι δεν είναι σαφές ακόμα τι χρονοδιάγραμμα θα θελήσει να ακολουθήσει το Συμβούλιο Αναμένεται όμως ότι ήδη από το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα βρίσκεται ε, στην ημερήσια διάταξη το πακέτο. Ε, δεν ξέρω βέβαια σε ποιο βαθμό θα θέλουν να έχουν καταλήξει σε κοινή θέση για τη δέσμη αυτή, αλλά ε, θα συζητηθεί σίγουρα και καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρξει τουλάχιστον μία γρήγορη παρουσίαση και να έχουμε τα σχέδια εκθέσεων. και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τα όσα έχουν ήδη κάνει ο Ντιόγκο Φέγιο και η κυρία Μπερέ. Αν δούμε σε γενικέ γραμμέ αυτή τη δέσμη, ε, με πιέζει και ο χρόνο βλέπω, διαπιστώνουμε ότι η ενίσχυση του Συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημιουργεί το εξή ερώτημα. Υπάρχει επαρκή ενίσχυση. Η οικονομική υποπτία στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά εδώ ε, αναφέρομαι κυρίως ε, στην πρόληψη, μας αρκεί, είναι αρκετά ισχυρή. Ε, φαντάζομαι ότι θα γίνουν και σχετικές συζητήσεις με το Συμβούλιο, αλλά είναι πολύ σημαντικό και εμεί ως Κοινοβούλιο να συνεχίσουμε και να πούμε ότι θέλουμε να έχουμε μια κοινή μέθοδο, να υπάρχει ε, και ισχυρό ρόλος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη δέσμη. Αυτό έχει ληφθεί υπόψη σε μεγάλο βαθμό για το θέμα των κυρώσεων, αλλά θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας απαντήσει και για το κατά πόσον τα κράτη-μέλη προχωρούν με καλό ρυθμό προς τους μεσοπρόθεσμους στόχους τους. Έχουν ληφθεί υπόψη αυτά, ε, υπάρχει αρκετό βάρος ε, και δεν είναι το Συμβούλιο αυτό που αποφασίζει, αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα σημαντικό επίση ερώτημα για το Κοινοβούλιο είναι πώς έχει ληφθεί υπόψη η δημοκρατική νομιμότητα. Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι θέλει να υπάρχει μια ισχυρή θέση, διότι εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη. Εμείς όμως, ή τουλάχιστον εγώ, θεωρώ ότι ελοχεύει ο εξή κίνδυνος ε, να πολιτικοποιηθούν πάρα πολύ τα θέματα και αυτό φυσικά δεν θα το θέλαμε σε καμία περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ισχυρός ρόλος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά η διαδικασία λήψη αποφάσεων και αξιολόγηση πώς γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα εποπτεύεται. Θα πρέπει να δούμε και τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος εξωτερικός παράγων που θα εξετάζει γενικώ το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβολίου, όχι αναπερίπτωση, αλλά περισσότερο Ε, πώς ε, ε, δίνουμε περισσότερο περιθώριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό φυσικά θα πρέπει να το εξετάσουμε σε επόμενες εβδομάδες και στους επόμενους μήνες. Τώρα, κάτι το οποίο σχετίζεται με τη συζήτηση και νομίζω ότι θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στις υπόλοιπες εκθέσεις, πώς θα ληφθεί υπόψη η εποπτεία του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν φορεί σε εθνικό επίπεδο που μπορούν να κάνουν την εποπτεία. Και μια ερώτηση επιπλέον, κατά πόσον θα πρέπει να αλλάξει το Σύμφωνο σταθερότητα και Ανάπτυξης και να γίνει μια εθνική πολιτική διαδικασία ή να περάσει ακόμα και στην εθνική νομοθεσία. Νομίζω ότι δεν έχω χρόνο. Ολοκληρώνοντας λοιπόν να πω ότι εγώ προσωπικώ, αλλά νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τους άλλους συζητητέ. είμαι στη διάθεσή σας και για σχόλια εδώ στη συνεδρίαση, αλλά και εκτός ε, συνεδρίασης, αν δεν φτάσει ο χρόνος, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιοδήποτε άλλου τρόπου, διότι νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ισχυρή θέση. Δεν ήθελα να σας διακόψω, διότι θέτατε κάποια ερωτήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα μέλη. Θα ήθελα όμως να ζητήσω από τους υπολείπους να προσπαθήσουν να τηρήσουν αυτά τα πέντε λεπτά, γιατί θέλω να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ομιλητές. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Φέιο, ο οποίος ασχολείται με την ε, ε, επιτάχυνση και τη διασαφήνιση εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ξεκινήσω τονίζοντας ότι το Κοινοβούλιο έχει μπροστά του ένα έργο αρκετά δύσκολο, αλλά απολύτως εφικτό να ολοκληρωθεί. Ήδη προσφάτως είδαμε ότι παρά τις ε, διαφορές σε διάφορα ζητήματα στη δέσμη εποπτείας καταφέραμε να προχωρήσουμε όπως και στην έκθεση για την οικονομική διακυβέρνηση. Έτσι λοιπόν και στο ιδέσμε για την οικονομική διακυβέρνηση, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια θέση κοινή και ισχυρή. Έτσι λοιπόν, αυτό θέλω να το τονίσω εδώ, παρά κάποιες, παρόλ, παρά κάποιες ε, αμέλειες, κάποιες διαφωνίες που έχουν προκύψει. Στην ε, Επιτροπή και στο Συμβούλιο δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία αμφιβολία για τη θέση που θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως και η πολιτική θέση μας θα πρέπει να είναι ενιαία και οι θέσεις που θα μας απασχολήσουν, συγκεκριμένα τέσσερις, ε, θα οδηγήσουν σε υποχρεωτικό σεβασμό της θέσης του Κοινοβουλίου λόγω της διαδικασία που ισχύει. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητηθούν αυτές οι εκθέσεις συνολικά ως δέσμοι, διότι είναι αλληλένδετες έχουν ε, να μας αποσχολήσουν ζητήματα τα οποία ε, έχουν πολλά κοινά σημεία. Έτσι λοιπόν, παρά τις διαφορετικές απόψεις, η πολιτική μας δέσμευση θα είναι καθοριστική εδώ. Είναι σημαντικό από πολιτικής άποψης και, και είναι ευαίσθητο το θέμα. Η έκθεση την οποία θέλω να σχολιάσω αφορά την τροποποίηση του κανονισμού 1467 ε, του 97 που θέλει να αποσαφηνίσει και να επιταχύνει τις διαδικασίες για το υπερβολικό έλλειμμα. Αυτός ο αρχικός κανονισμός του 1997 αναθεωρήθηκε το 2005. Τώρα βρισκόμαστε στη νέα αναθεώρηση. Η όλη η συζήτηση έχει ήδη πάρει κάποιες κατευθύνσεις και οι αλλαγές που προτείνονται, θέλω να ενημερώσω σχετικά τους συναδέλφους, έχουν διαφορετικό, διαφορετικές ε, Κάποιες τεχνικές, ε, διαδικαστικές, έχουν σχέση με την ύπαρξη, την θέση σε ισχύ της νέας συνθήκης. Άλλες είναι επί της ουσίας. Επί της ουσίας αλλαγές έχουν να κάνουν κυρίως με το θέμα της υλοποίησης του κανονισμού αυτό όχι μόνο για τις περιπτώσεις ελλείμματος, αλλά και του δημοσίου χρέους. Υπάρχει μια ε, συνιστόσα λοιπόν διορθωτική του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης προκειμένου να ε, αποφευθούν τα σοβαρά σφάλματα στις πολιτικές προπολογισμού των κρατών μελών. Δηλαδή θα πρέπει να εφαρμόζεται το σύστημα αυτό και στο δημόσιο χρέος και στα όρια του. Από την άλλη προβλέπονται και αλλαγές σε σχέση με την καλύτερη ενημέρωση από τα κράτη για την εξέλιξη του χρέους τους. Ήθελα εδώ να τονίσω ότι σύμφωνα με την πρόταση τα κράτη-μέλη που ξεπερνούν το 7% στο ΑΕΠ θα πρέπει να λάβουν ε, μέτρα για, την, ε, ε, για το μετριασμό του χρέους καθώς και ετήσια μέτρα ώστε σε μία τριετία να μπορέσουν να μην ξεπερνούν το κατόφλι αυτό του 7%. Επίσης η εξέλιξη του δημοσίου χρέους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις ε, φάσεις της διαδικασίας για το δημόσιο έλλειμμα. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί λοιπόν μία εξέταση και να έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην αύξηση του χρέους. Επίσης η ονομαστική αξία της Αύξηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη καθώς και η σχετική κίνδυνη με την ε, δομή του χρέου. Θα πρέπει εδώ να θέσω ένα ερώτημα που θα ήταν καλό να μα αποσχολήσει στη συζήτησή μα. Θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη πειθαρχία σε όλα αυτά τα ζητήματα και στο πώ αντιμετωπίζονται και το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να δει τι κατευθύνσει πρέπει να δοθούν ε, για τι ε, δημόσιε αυτέ πολιτικέ που είναι κινητήριο δύναμη τη ανάπτυξη. Ιδίω το σκέλος ε, της Ανάπτυξη είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε διτέρως κύριε Φέιο. Και τώρα έχουμε την κυρία Φερέιρα, η οποία θα μας μιλήσει για την πρόληψη και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι που προηγήθηκαν ήδη ανέφεραν τη σημασία Τη προβολή που πρέπει να δώσουμε στη δέσμη αυτή, στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όχι μόνο το θεσμικό ρόλο του Κοινοβουλίου, αλλά και στην ε, ιδιαίτερη αρμοδιότητα, την νομική αρμοδιότητα, το νομικό κύρος που έχει πλέον το Κοινοβούλιο να, ως συνομοθέτης. Είναι λοιπόν σημαντικό δημοσίως ο ρόλος, ο νέος αυτός ρόλος να καταστεί σαφής. Όσα συζητούμε δεν θα μπορέσουν να περατωθούν χωρίς τη δική μας τη συμβολή του Κοινοβουλίου. Θέλω λοιπόν να τονίσω, όπως έκαναν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, το ενδιαφέρον που έχουμε για αυτό το θέμα, όπως και για παλιότερα θέματα. Και εδώ είναι σημαντικό να έχουμε μια ισχυρή και ενιαία θέση ως Κοινοβούλιο, ανεξαρτήτως των ε, διαφορών των πολιτικών που υπάρχουν προφανώς ε, μεταξύ των παρατάξεων. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση για άλλη μια φορά να καταλήξουμε σε μια ενιαία θέση ισχυρή ώστε να επειρασπιστούμε τα συμφέροντα και της Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών. Πέραν αυτών και σε σχέση με την εν λόγω έκθεση, την νομική πράξη για την οποία έχω αναλάβει δηλαδή η συγγήτρια, η έκθεση αυτή συνδέεται άμεσα με, άλλη, με τις άλλες εκθέσεις που αποτελούν μέρος της δέσμης για την χρηματοοικονομική διακυβέρνηση. Είναι τα νομικά μέτρα για να διορθωθούν οι μακρονομικές ανισορροπίες στην Ευρωζώνη. Εδώ η συγητής είναι ο συνάδελφος Χάγκλουντ. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε την παρακολούθηση και διόρθωση των μακροοικονομικών ισορροπιών από κοινού με το σύστημα κυρώσεων. Το σύστημα κυρώσεων που ακριβώς προβλέπει η έκθεση του Καρλ Χάγκλουντ. Η διάσταση αυτή είναι μια διάσταση τελείως καινούρια. Εδώ διαφέρει και όλα η έκθεση αυτή σε σχέση με όσα παρουσίασε ο συνάδελφο Διόγκου Φέγιο, σε σχέση με το Σύμφωνο ανάπτυξης και σταθερότητας Το σύμφωνο αυτό το έχει υποστεί αρκετές αναθεωρήσεις και τώρα διευρύνεται. Καλύπτει και τον έλεγχο του χρέους και τις κυρώσεις που μπορεί να σχετίζονται με το χρέος. Όμως στη δική μου την έκθεση, στην εν λόγω έκθεση, αυτό που διακυβεύεται είναι η παρατήρηση των μακροοικονομικών ισορροπιών στις οικονομίες των χωρών και μετά με την έκθεση του κ. Χάγκλουντ ε, θα περάσουμε και στη διάσταση των κυρώσεων για τις ίδιες ακριβώς ανισορροπίες. Ως τώρα, η κατάσταση την οποία έχουμε γνωρίσει είναι να έχουμε πολλές συστάσεις που προκύπτουν από διαφορετικές πηγές των διαφορετικών των θεσμικών οργάνων που κάποιες φορές προσκαλούν οι γενικές οικονομικές γραμμές, broad economic guidelines, να προσαρμόζονται. Από το 2008 η ομάδα της Ευρωζώνης ξεκίνησε μια διαδικασία συστηματικής παρακολούθησης της ανταγωνιστικότητας εντός της Ευρωζώνης και το 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να γίνει πιο αποτελεσματική ακόμη η παρακολούθηση των διαφόρων τάσεων και εντάσεων. Το Κοινοβούλιο και με την έκθεση Φέγιο και με την έκθεση Μπερές έχει ασχοληθεί με το ευρύτερο αυτό θέμα της μακροοικονομικής ανισορροπίας. Ζήτησε το Κοινοβούλιο να γίνει μια πιο συστηματική δουλειά για την εξέταση των αιτίων των μακροοικονομικών ανισορροπιών και να ληφθούν υπόψη οι πτυχές ανάπτυξης της απασχόλησης, της ανεργίας, οι, πραγματι... οι μεταβλητές οι πραγματικές καθώς και οι μεταβλητές οικονομικές ονομαστικής αξίας πως τώρα δεν είχαν ληφθεί, υπόψη. Αυτές είναι οι δύο βασικές ε, πτυχές που ανέπτυξαν οι εκθέσεις Φέγιο και Εμπερές. Εδώ τώρα στη σύνταξη αυτής της έκθεσης θα ασχοληθούμε από τη μια με την διασάφηση αυτών που θεωρούμε πραγματικές ε, μακροοικονομικές ανισορροπίες, καθώς μας λέει η Επιτροπή ότι θα αναβάλει για ένα μεταγενέστερο στάδιο τον ακριβή ορισμό του τι σημαίνει μακροοικονομική ανισορροπία. Μιλά για μια δημιουργία ενός scoreboard, ενός ε, πίνακα δηλαδή που θα συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένους δείκτες, όμως δεν μας λέει ποιοι θα είναι αυτοί οι δείκτες. Το Κοινοβούλιο σε διάφορες περιπτώσεις ζήτησε οι δείκτες αυτοί ε, να είναι οι δείκτες ανάπτυξης, απασχόλησης, ανεργίας, ένδυας και το καθεξής, ενώ από την άλλη η Επιτροπή αφήνει για αργότερα τον κατάλογο με τους δείκτες που θα καλύπτονται μελλοντικά. Νομίζω ότι το ζήτημα αυτό είναι αποφασιστική σημασία. Θα πρέπει να το θίξουμε ως ε, Κοινοβούλιο. Και αυτό καθώς και την ταχεία μετάβαση προς ένα κατάλογο επιπλέον κυρώσεων, χωρίς να έχει ετοιμαστεί ο άλλος κατάλογος ε, αναγκαστικά προηγουμένως. Γιατί και σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να έχει ετοιμαστεί και, και αυτός ο κατάλογος προκειμένου να, είναι, να υπάρχει συνέπεια στην όλη δέσμη της ε, οικονομικής διακυβέρνησης. Το ζήτημα λοιπόν των κυρώσεων ούτως ή άλλως νομίζω θα το θίξει και ο συνάδελφος Χάγκλουντ. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκουλάρ, έχετε το λόγο για την ουσιαστική ενίσχυση της μονοσομενικής εποπτείας στη ζώρη του ευρώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό που μπορούμε σήμερα το πρωί να έχουμε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους ευρωβουλευτές, πέραν δηλαδή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, και έχει επιπτώσεις και για τους πολίτες και για τις αγορές. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση λοιπόν να αποτύχουμε στην αποστολή μας για τη βελτίωση του συστήματος. Οι προτάσεις της Επιτροπής, καταρχήν θα ήθελα να πω, ακολουθούν μια σωστή κατεύθυνση. Έγινε μια καλή επεξεργασία του θέματος, αφορά την πειθαρχία. Έχει δίκιο η Επιτροπή όταν λέει ότι πρέπει να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, λιγότερη δυνατότητα διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών και βεβαίως να συμπεριλάβουμε και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έχει γίνει ήδη μια συγκεκριμένη εργασία. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Όταν δημιουργήθηκε το ευρώ, δεν θεωρήσαμε ότι το σύστημα αυτό θα διαρκούσε. Ήταν μια μεταβατική περίοδος και τα κράτη σήμερα, οι κυβερνήσεις, θεωρούν ότι αυτό θα πρέπει να διαρκέσει. Αυτό είναι ορθό ή όχι. Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε και να σκεφτόμαστε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο in the box, είτε θα ανοίξουμε ε, τις δυνατότητες και θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τις εξωτερικές επιπτώσεις. Αυτό λοιπόν που σήμερα μας αφορά είναι ο συντονισμός σε εθνικό επίπεδο της οικονομικής πολιτικής και να δούμε αν οι αποφάσεις βασίζονται σε ένα αυτόματο σύστημα λήψης αποφάσεων είτε σε μία απόφαση που λαμβάνεται μετά από σκέψη και το ερώτημα είναι εδώ αν θα συνεχίσουμε να παίρνουμε τις αποφάσεις με αυτόν τον τρόπο. Ο συντονισμός, κατά την άποψή μου, προϋποθέτει αυτοματισμό. Και ο αυτοματισμός δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το σύστημα θα λειτουργεί από μόνο του και θα λαμβάνονται αποφάσεις που οδηγούν σε κυρώσεις. Η επιθυμία μας δεν είναι η αύξηση των κυρώσεων, αλλά ο συντονισμός προϋποθέτει σαφώς και περισσότερο αυτοματισμό, περισσότερες αρμοδιότητες στην Επιτροπή για μια ανάλυση η οποία θα βασίζεται σε αυτήν την δυνατότητα συντονισμού. Τώρα, ο δημοκρατικός έλεγχος των αποφάσεων. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε περισσότερο αυτοματισμό, περισσότερη πειθαρχία. Κάτι το οποίο βεβαίως μας οδηγεί σε κάποιες πολιτικές αποφάσεις, επιλογές. Θα πρέπει να ελέγξουμε λοιπόν τη δημοκρατική νομιμότητα. Σήμερα και τις επόμενες ε, εβδομάδες, όπως είπε και η Ελίζα, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες, τους δημοσιογράφους, ότι δεν υπάρχει μία task force η οποία και κλεισμένων των θυρών αποφασίζει, ότι δεν υπάρχει η συνάντηση της Ντοβίλ με δύο επικεφαλής κρατών οι οποίοι αποφασίζουν. Υπάρχει ένα κοινοβούλιο που εκπροσωπεί όλες τις πολιτικές ευαισθησίες, όλες τις πολιτικές και εθνικές απόψεις. Υπάρχει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και πιο μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι θα πρέπει σε αυτές τις διαδικασίες να συμπεριλάβουμε περισσότερη δημόσια συζήτηση. Οι προτάσει τη Επιτροπή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θα πρέπει ίσω λοιπόν να υπάρξει και μια φάση ακροάσεων, συζητήσεων. Όλα αυτά τα λέω χωρίς να έχω απολύτως καμία προκαθορισμένη άποψη. Ίσως όμως θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να μπορούν να υπερασπιστούν τις απόψεις τους και να υπάρξει μια συζήτηση δημόσια, διασυνοριακή, διακρατική και να μην αφήσουμε τον τύπο, ιδιαίτερα τον λαϊκιστικό τύπο, να κάνει εδώ κάποιες ε, δηλώσεις. Αν θυμάστε την Άνοιξη ακούσαμε τον κύριο Παπανδρέου, ακούσαμε την ενδιαφερόμενη χώρα να προωθήσει τις απόψεις της. Αυτό είναι μια δημοκρατική διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί, αλλιώς κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου οι λαϊκιστικές τάσεις θα υπερισχύσουν και θα επικρατήσει η άποψη ότι οι Βρυξέλλες ε, επιβάλλουν ε, κάποιες αποφάσεις. Η Επιτροπή προτείνει εδώ να αντιστρέψει την πλειοψηφία, δηλαδή με ενισχυμένη πλειοψηφία να μπορεί να απορριφθεί μια πρόταση. Εδώ όμως θα χρειάζεται μια προεργασία νομοθετικού τύπου. Η Ελίζα μίλησε για τους καλούς μακροοικονομικούς δείκτες. Και αυτό χρειάζεται έναν σχεδιασμό, ο οποίος θα πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί οι κυρώσεις ανέρχονται στο 0,2 του ΑΕΠ. Γιατί, πώς το επιλέξαμε αυτό το 0,2 του ΑΕΠ. Δεν έχω άποψη από αυτού. Κάτι άλλο, η στρατηγική για το 2020 θα πρέπει να δούμε το θέμα της πειθαρχία και το θέμα της θετικής ε, προσέγγισης της ανάπτυξης δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Ζητώ λοιπόν να ενημερώσουμε και τους πολίτες και τις αγορές έτσι ώστε το προϊόν που θα αναπτύξουμε να έχει αξιοπιστία. Θα σε ευχαριστώ. Θα περάσουμε στην έκθεση του κυρίου Χάγκλαντ. Πρόκειται για τα μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι είμαι θετικά διακείμενο στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε, μια φιλόδεξη δέσμη ε, για να συζητήσουμε. Βέβαια, θα μπορούσαμε κάλλιστα να δαπανίσουμε αρκετό χρόνο και να συζητάμε το πώς θα αντιμετωπίσει το Συμβούλιο αυτό ε, είναι καλό το γεγονός ότι έχουμε ένα φιλόδοξο πακέτο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται το Συμβούλιο και με τον τρόπο με τον οποίο κάποια κράτη-μέλη κάνουν συμφωνίες ε, με ανησυχεί γιατί δεν ξέρω σε τι διαπραγματευτική θέση θα βρισκόμαστε σε κάποιους μήνες. Είναι επίση σημαντικό να έχουμε και εμεί ω Κοινοβούλιο μια φιλόδοξη προσέγγιση, αλλά να είμαστε όσο το δυνατόν ενωμένοι. Γιατί αν δεν υπάρχει ευρεία συνένεση, ε, και δεν υποστηρίζει τη γραμμή του Κοινοβουλίου, θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο και να καταλήξουμε σε τελική θέση. Επίσης, μεγάλη πρόκληση αποτελεί και το σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Όπως είπε και η Ελίζα, κατά πάσα πιθανότητα ο κάθε ευρωβουλευτής έχει δική του άποψη για το πακέτο αυτό, που σημαίνει ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση διότι ναι μεν για τα οικονομικά θέματα δεν ενδιαφέρονται οι περισσότεροι ευρωβουλευτέ, αλλά φαντάζομαι ότι για αυτή τη δέσμη νομοθετικών μέτρων θα έχουν όλοι άποψη. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ακούσουμε την άποψη όλων και να συμφωνήσουμε όλοι από κοινού για το τι ακριβώς θέλει το Κοινοβούλιο για το πακέτο αυτό. Όταν ξεκινάει η ανάλυση και το πιο σημαντικό είναι να αναλύσουμε ποια είναι η εναλλακτική λύση στο να ακολουθήσουμε απλώς την ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι έχουμε ένα φιλόδοξο πακέτο και ακολουθείται μια διαφορετική οδός και θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι ακριβώς κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πολύ αυστηρή θέση επί του θέματος και νομίζω ότι οι πολίτες της Ευρώπης, κυρίως ε, οι χώρες Ευρωζώνης, περιμένουν από εμά κάτι φιλόδοξο. Θα πρέπει να δείξουμε λοιπόν και στους πολίτες αλλά και στις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να κάνουμε κάτι, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και μια στεναρή θέση. Για να επιτευχθεί βέβαια αυτό θα πρέπει να έχουμε μια ε, καλή ε, συζήτηση. Χαίρομαι που είχαμε δύο πολύ καλές συνεδριάσεις με τους εισηγητές, έγινε μια πολύ καλή πρώτη συζήτηση, αυτή είναι σωστή προσέγγιση και νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να διαμορφώσουμε μια καλή θέση ως κοινοβούλιο. Ένα θέμα το οποίο επίσης θα αποτελέσει πρόκληση είναι το γεγονός ότι πολλοί εθνικοί πολιτικοί και βουλευτές έχουν ε, στεναρές θέσεις επί του θέματος, το οποίο ναι μένει είναι καλό, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει και κάποιες πιέσεις. Και επίσης το γεγονός ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις νομικές πτυχές. Ε, άκουσα και κάποιες παρατηρήσεις για κάποιους που θέλουν να τονίσουν ότι η, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν συνάδει με όλες τις συνθήκες. Εγώ δεν είμαι πυρογνώμων επί των συνθήκων, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τα αναλύσουμε αυτά τα θέματα και να είμαστε βέβαιοι ότι όλα συνάδουν με τις ε, κείμενες συνθήκες. Κάποιοι βέβαια έφτασαν και λίγο πέρα από τα όρια και πρότειναν και αλλαγέ των συνθήκων, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό αφορά το πακέτο μας. Εν κατακλείδη, όσον αφορά την όλη δέσμη, νομίζω ότι εξαρτώμεθα ο ένας από τον άλλον. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου χωρίς να γνωρίζω τι κάνει η κυρία Φερέιρα και νομίζω ότι αυτό λειτουργεί και αντίστροφα. Θα πρέπει αυτά τα οποία προτείνουμε, οι κυρώσει που προτείνουμε, συνάδουν και με τα όσα έχουμε στην όλη δέσμη και να έχουμε μια συνολική προσέγγιση. Θα πρέπει δηλαδή να βρούμε και μία θέση για τους δείκτες και για κάποια θέματα για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και εδώ συμφωνώ με τα όσα είπε και η κυρία Φερέιρα. Ακόμα δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς μιλάμε και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μας ε, στο πακέτο. Να είμαστε βέβαιοι ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα όλοι, διότι και από άλλες εκθέσεις που έχουμε συζητήσει εδώ στην Επιτροπή ε, φαίνεται ότι δεν συμφωνούμε όλοι ως προς ένα κοινό ορισμό για το τι ακριβώς σημαίνει οικονομική ανισορροπία. Ε, νομίζω ότι αν εργαστούμε ε, όλοι μαζί από κοινού θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό πακέτο και θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση για το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τέλος η κυρία Φόρντ, η οποία είναι η συγγήτρια για τις απαιτήσει για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή αποτελεί ουσιαστικά το εφαλτήριο για όλα τα υπόλοιπα, διότι είναι η έκθεση από την οποία ζητούμε από τα κράτη-μέλη να μας δώσουν στοιχεία, ε, να ετοιμάσουν στοιχεία και να τα δώσουν στους ε, γείτονές τους και στο ευρύ κοινό και νομίζω ότι αυτό αποτελεί το ένασμα για όλες τις υπόλοιπες συζητήσεις και επομένως θα πρέπει να έχουμε ακριβή και προσβάσιμα δεδομένα, πιο ακριβή και πιο προσβάσιμα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν για να μην καταλήξουμε στη σημερινή κατάσταση. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να βελτιωθεί το επίπεδο των δημόσιων ε, δεδομένων και όπως πολύ ε, συχνά λέμε στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ρίξουμε φως ε, στην υπόθεση γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε περισσότερη διαφάνεια. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην πρότασή της προσθέτει πολλές πληροφορίες που θα ήθελαν να δώσουν επιπλέον. Παραδείγματο χάρη ε, τα θέματα της ευθύνης. Εμείς εδώ στην ΟΜΑΝΑ πολλές φορές λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες ε, πληροφορίες. Επίσης, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν εθνικές διαφορές μεταξύ των χωρών και δεν θα μπορούμε να έχουμε μία ενιαία προσέγγιση για όλες τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Η ομάδα ειδικών καθηκόντων Φανερόμπα που ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά διεξοδικά ακολούθησαν μια δυτική προσέγγιση. Υπάρχει ένα ελάχιστο ε, πακέτο δεδομένων που θα πρέπει να δίνουν τα κράτη-μέλη, κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις και μετά από εκεί και πέρα ίσως θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες ε, μη δεσμευτικέ ε, απαιτήσεις τις οποίες θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη. Και εδώ νομίζω ότι έχουμε κάτι χρήσιμο. Θα μπορούσαμε ίσως να δούμε λίγο καλύτερα γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η δυτή προσέγγιση και γιατί η Task Force θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η δυτή προσέγγιση. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο αναφέραμε στην έκθεση ΦΕΙΟ είναι ότι θα πρέπει να έχουμε δύο τρόπους εποπτείας. Ένα τρόπο όταν ε, όλα πηγαίνουν καλά, αλλά όταν υπάρχουν προβλήματα να μπορούμε να εξετάσουμε λίγο περισσότερο τα πράγματα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι υπόλοιποι ε, όταν φτάνουν σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο εποπτείας εξετάζουν αυτά. Ο Τζόρτζ Μπερναρσό είπε ότι αν μαζέψουμε όλους τους οικονομολόγους στον κόσμο και ακούσουμε την άποψή τους και πάλι δεν θα έχουμε μια σαφή θέση για τίποτα. Ε, είναι λοιπόν αυτό ο οποίο είναι ο πλέον αρμόδιο για να λάβει αποφάσει για τα κράτη-μέλη. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ε, ή οποιοδήποτε άλλο ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι φορείς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτό το ενισχυμένο επίπεδο εποπτείας Ορισμένε φορέ όταν τα κράτη-μέλη καταρτίζουν τον προπολογισμό του μπορεί να μην θεωρούν ότι θα πρέπει να συμπίπτουν μετά όσα ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθούν με να ακολουθήσουν την άγουσα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής αλλά να εξηγούν πότε ε, ξεφεύγουν και γιατί. Αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο στο κείμενο. Κάτι επίση σημαντικό που θα πρέπει να δώσουμε στο ευρύ κοινό είναι το γεγονός ότι ζητάμε από τα κράτη-μέλη να να έχουν προβλέψεις για τον προπολογισμό τους με διάφανο και διεξοδικό τρόπο και θα πρέπει να κάνει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δικά της στοιχεία. Ε, διότι κάποιο δεν μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει πού πάει ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όταν έχουμε μία τριετή πρόβλεψη. Και επειδή ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μεγαλύτερο από τουλάχιστον ε, ε, τα μισά κράτη-μέλη, θα πρέπει να προσέχουμε λίγο καλύτερα τι κάνουμε κι εμείς. Ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε στην ε, ομάδα μου είναι κατά πόσον ε, είναι αποτελεσματικές αυτές οι, κυρές, οι κυρώσεις και αν δεν είναι αποτελεσματικές υπάρχει ίσως η ανάγκη να υπάρχει κάποιος τρόπος επίλυσης κρίσεων που να θεωρείται αξιόπιστος. Αυτό Ε, η έννοια που λέμε ότι η αγορά θα πρέπει να ε, αντιμετωπίζει, να αναλαμβάνει κάποιο βάρος της ευθύνης, ε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποδεκτή, δεν ξέρω αν ο φορολογούμενος είναι αυτός που πρέπει να πληρώνει πάντα. Θα πρέπει να βλέπουμε και τι γίνεται να υπάρχει μια προσέγγιση που θα έχει ως βάση την αγορά. Θεωρώ ότι αυτές οι έξι νομοθετικές προτάσεις είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον. Ευχαριστώ. Για να μπορέσουμε να διαρθρώσουμε λίγο κάπως τη συζήτηση και να είναι τα πράγματα όσο πιο απλά γίνεται. Έχω κάποιους όδης εισηγητές που είναι και εισηγητές και έχουν ήδη μιλήσει, αλλά θα κάνουμε το εξή. Εάν ε, κάποιο όδης έχει ζητήσει να μιλήσει, θα του δώσουμε το λόγο. Μέχρι τούδε μόνο τρει έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριο Λάγκεν έχει πάντα καλύτερη ιδέα από την πρόεδρο. Θα σημειώσω λοιπόν τους κοιόδης, θα τους προσθέσω στο κατάλογο των ομιλητών. Έχω και τρεις ε, συναδέλφους που δεν είναι σκιώδης εισηγητές, αλλά φυσικά θέλουν το λόγο και θα τους τον δώσουμε. Αν είστε σκιώδης εισηγητής για κάποια έκθεση και θέλετε να κάνετε μια παρατήρηση στον εισηγητή, να απευθύνετε την ερώτηση αυτών ή την παρατήρηση αυτών για να μπορέσει να το λάβει υπόψη. Να δω πώς θα ξεκινήσουμε γιατί είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Ο κύριος Γκυγκόλ θέλει να μιλήσει πρώτο για ένα λεπτό. Για δύο λεπτό, είπα θα δώσω στους κοιότης το λόγο. Κύριε Γκίγκολτ, έχετε το λόγο. Ή αν δεν θέλετε να μιλήσετε και θέλετε να δώσετε το χρόνο σας στον κύριο Λάμπερτ. Εκτός μικροφώνου το σχόλιο. Η ε, πρόεδρος, πρώτα θα ακούσουμε τους σκιώδεις συγητές. Δεν είστε στον κατάλογο. Αλλάξαμε τον κατάλογο. Εγώ είμαι σκιώδης συγητής και για τις έξι εκθέσεις. Δεν σας έχω στον κατάλογο, λέει η πρόεδρος. Ωραία. Ξεκινάτε εσείς κύριε Λάμπερτς για να μην ε, μακρηγορούμε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εντυπωσιάστηκα, ξαφνιάστηκα από την έλλειψη στάση επικοδομητικής από μέρους του Συμβουλίου. Δεν θα ξεκινήσω τώρα ένα θεσμικό, μια θεσμική αντιπαράθεση, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά αν θέλουμε να ακουστούμε θα πρέπει να δείξουμε συνοχή και αυτό έγινε με την έκθεση Φέγιο. Πιστεύω ότι όλοι οι εισηγητές μας έδειξαν ότι πρέπει να πάμε προς αυτή την κατάθεση. Οι πράσινοι λοιπόν θέλουν να ακολουθηθεί αυτή η κατεύθυνση. Πρόκειται για θέματα πολιτικά και βεβαίως υπάρχει δυνατότητα εδώ μεγάλη να διαιρεθούμε. Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά όλοι να προσπαθήσουμε να μην πέσουμε σε αυτήν την παγίδα και να οδηγηθούμε σε επικοδομητικές προτάσεις. Τρία σχόλια όσον αφορά το πακέτο προτάσεων. Πρώτον, αν θέλουμε να τηρηθούν κανόνες, χρειάζονται κυρώσεις. Αυτό είναι κάτι που δεν το αμφισβητεί κανείς. Χρειάζεται να αποφασίσουμε, να στηρίξουμε έξυπνους κανόνες. Και σαφώς σήμερα οι κανόνες δεν ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη. Κοιτάξτε τους κανόνες που αφορούν τα ελλείμματα. 100% του ΑΕΠ για κάποιες χώρες. Οι κανόνες προτείνουν σήμερα στις χώρες αυτές να υπάρξει ένα πλεόνασμα της τάξης του 5% κάθε χρόνο, 5% συν στο ΕΠ, έτσι ώστε να ε, υπάρξει εξισορρόπηση. Αυτό είναι κάτι το ρεαλιστικό. Τι άλλο μπορούμε να προτείνουμε έτσι ώστε να υπάρξει σύγκληση. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο επιμένει ότι πρέπει να υπάρξει μία προσέγγιση, τιμωρία, κύρωση και θετικό κίνητρο. Εμείς βλέπουμε όμως στις προτάσεις αυτές να υπάρχει απλώς μία πολιτική κυρώσεων και όχι θετικών κινήτρων. Θέλουμε δηλαδή να δώσουμε στα κράτη την ε, δυνατότητα να δουν και την θετική πλευρά, το θετικό κίνητρο για να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το σημείο. Τρίτη παρατήρηση. Η Επιτροπή μας απογοήτευσε ως ένα βαθμό, κοιτώντας τις ε, δηλώσεις του Επιτρόπου Ολιρέν την Άνοιξη, καταλάβαμε ότι είχε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν μακροοικονομικές ανισορροπίες και ότι θα έδινε έμφαση σε κάποιους δείκτες οι οποίοι να είναι εφικτοί ως προς την υλοποίησή τους. Εδώ βλέπουμε όμως ότι υποχωρεί σε κάποια σημεία. Λέει θα δούμε, θα το ξανασκεφτούμε και θα κάνουμε προτάσεις. Και οι προτάσεις τελικά φαίνεται να γίνονται μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου, χωρίς λόγος να δίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε λοιπόν εδώ να διασφαλίσουμε ότι εξετάζονται τα σωστά σημεία. Όχι δηλαδή μόνο τα δημόσια ελλείμματα, αλλά και τα ελλείμματα στον ιδιωτικό τομέα και ισορροπίες, εξάρτηση από αρνητικό περιβάλλον. Όπως είπε και η Σιλβή, το θέμα του κινδύνου της απειλής να μην κατανοήσουν οι πολίτες, να χάσουμε δηλαδή την στήριξη των πολιτών. Και πιστεύω ότι οι επιθέσεις που γίνονται εδώ δεν γίνονται μόνο από τα λαϊκιστικά κόμματα ή εφημερίδες, αλλά και από συγκεκριμένα κράτη. Θα πρέπει λοιπόν για να κάνουμε κάτι και να προχωρήσουμε σε κάτι, να έχουμε την συμμετοχή του Κοινοβουλίου, όχι μόνο στο νομοθετικό κομμάτι, σε όλη τη διαδικασία και στο εκτελεστικό. Χρειαζόμαστε διαφάνεια και μόνο μέσω διαφάνειας μπορούν να συμμετάσχουν και οι πολίτες. Και την ίδια ώρα θα πρέπει τα κράτη-μέλη να καταλάβουν ότι δεν μπορούν και κλεισμένων των θυρών και στις ε, συνεδριάσεις του Συμβουλίου να λένε Α και όταν βγαίνουν να λένε Β. Σιλβί, συμφωνώ μαζί σου. Πρέπει να βρούμε εδώ το θετικό κομμάτι της στρατηγικής του 2020 και το αρνητικό κομμάτι των κυρώσεων. Ξεπέρασα το χρόνο μου, αλλά νομίζω ότι πραγματικά είμαι σκιώδης για όλες τις εκθέσεις. Πρόεδρος, κύριε Λάγκεν, θέλετε να προεδρεύσετε στη θέση μου. Αν θέλετε, λάτε εδώ και πάτε θέση. Ο κύριος Λάμπερτς είχε το λόγο πιο πολύ, γιατί ήταν σκιώδης για έξι εκθέσεις. Τελείωσα εξάλλου. Λοιπόν, θα διαβάσω τον κατάλογο των ομιλητών. Madam Hubner, Mr. Giegold, Mrs. Swinburne, Mr. Handel, Mr. and Mr. Juan Όλοι είναι σκιώδες εισηγητής, όλοι αυτοί και ο κύριος Σμιτ, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής, έχετε το δικαίωμα να πάρετε το λόγο, όπως και η κυρία Λούλινγκ. Λοιπόν, όλοι θα μπείτε στον κατάλογο, θα το προσπαθήσουμε, αλλά πρώτα θα πάρουν το λόγο οι οι συγητές, οι Και καταλαβαίνετε ότι αν μιλήσετε περισσότερο χρόνο, μειώνουμε το χρόνο των εισηγητών στο τέλος. Αλλά ο κύριος Λάμπερτς είχε δικαίωμα να μιλήσει παραπάνω γιατί ήταν σκιώδης για έξι εκθέσεις. Like my Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με την ε, απογοήτευση που εξέφρασαν και άλλοι συνάδελφοι για το πού θέλει να πάει το Συμβούλιο με την ανακοίνωσή του, διότι φυσικά δεν βοηθά τη συζήτηση όλο αυτό. Συμφωνώ επίσης και με τη δεύτερη παρατήρηση, μια κάποια έκπληξη που έχουμε όλοι για το θέμα. Δεν θα πρέπει να βιαστούμε, θα πρέπει να ακούσουμε, να ακούσουμε τι έχει να πει ο λαός, οι εμπειρογνώμονες, να ακούσουμε το ευρύ κοινό, διότι πρέπει να γνωρίσουμε περισσότερα. δεν μπορούμε να ακούσουμε μόνο μία άποψη επειδή κάτι είναι πήγον. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι οι κανόνες και οι κυρώσεις μπορούν να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Φυσικά αν υπάρχει νόημα στους κανόνες. Καταρχάς, Ευρωζώνη. Είχαμε συμφωνήσει ότι τα κριτήρια κοινού νομίσματος δεν τηρούνται στην Ευρωζώνη, όπως ε, γίνεται στις ΗΠΑ... Γι' αυτό ακριβώς και δημιουργήσαμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και περιμέναμε τα κράτη-μέλη να επιδείξουν μια κάποια σοφροσύνη Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε κάποιο να τι αποκολώσει κυρώσει, αλλά το γεγονό ότι όταν ε, κάποιε χώρε κάναν αίτηση να ενταχθούν στην Ευρωζώνη και πέρασαν και από μία διετή περίοδο δοκιμαστική, έπρεπε στο τέλο αυτή τη περίοδου να περάσουν τι εξετάσει, αν θέλετε. Αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν κύρωση. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτή τη γραμμή, δεν είστε επιλέξιμο. Και φυσικά κάποιος θα περίμενε ότι αυτό το οποίο απέκτησε σε διάρκεια αυτής της ε, δοκιμαστικής διετής περίοδου να συνεχιστεί. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε τι θα μπορούσε να συμβεί η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση με όλες αυτές τις ε, λύσεις οι οποίες ε, δόθηκαν, τα πακέτα διάσωσης και υποστήριξης. Και τώρα περνάμε από το δοκιμαστικό στάδιο και ε, εξετάζουμε τι συνέβη μετά από ένα γεγονός. Τι συνέβη αυτό για πολλές χώρες. Ε, τεράστια χρέη για τους λόγους που αναφέθηκαν, ε, πακέτα υποστήριξης και λύσεις οι οποίες ελήφθησαν. Τι σημαίνει όμως αυτό για τις διαρθρωτικές αλλαγές. Μιλάμε για την περίοδο μετά από ένα ε, πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο δεν είχε συμβεί για πάρα πολλά χρόνια. Θα πρέπει κάποιος λοιπόν να μας εξηγήσει γιατί λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο όλες αυτές οι περίεργες ε, μέθοδοι που ακολουθούμε. Και φυσικά θα πρέπει να εφαρμοστούν σε χώρες που όπως σας είπα έχουν τεράστια δημόσια χρέη λόγω των τακτικών που ακολούθησαν. Νομίζω ότι αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να κάνω πιο γενικά σχόλια σε όλες μας τις ε, χώρες έχουμε διαφορετικές ε, συνθήκες ε, δημοσιονομικές, μακροοικονομικές για την ρύθμιση των ελλημάτων παραγωγή, τους δείκτες παραγωγικότητας, τις εμπορικές συναλλαγές και όντως η αντιμετώπιση τους μπορεί να είναι κοινή, αλλά τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Κάτι που θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε σε όλους τους πολιτικούς είναι ότι χρειάζεται σαφήνεια και για τους πολίτες της Ευρώπης, αλλά και για τις χρηματαγορές. Γιατί βλέπουμε ότι όταν διστάζουν οι πολιτικοί για τους πολίτες τα πράγματα δεν είναι σαφή και για τις χρηματαγορές ε, βλέπουμε έντονες διακυμάνσεις με επιπτώσεις στα ελλείμματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε σαφή κατεύθυνση όταν μιλάμε παραδείγματος χάρη για τις κυρώσεις. Και θα πρέπει οι κυρώσεις αυτές να είναι πραγματικές κυρώσεις έτσι ώστε σιγά σιγά να ανακτήσουμε και την εμπιστοσύνη των αγορών αλλά και της, την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η χώρα μου η Λετωνία, η οποία χτυπήθηκε από την κρίση, γνώρισε αυτήν την κατάσταση και πάντα ο Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση εξηγούσαν στον κόσμο πού ήταν οι δυσκολίες και ότι ήταν απαραίτητο ένα σχέδιο λιτότητας για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Σαν αποτέλεσμα είδαμε ότι όχι μόνο υλοποιήθηκαν αυτά τα μέτρα λιτότητας, όχι μόνο η οικονομία μας σήμερα πάει καλύτερα, αλλά η πλειοψηφία των πολιτών μας στήριξαν αυτήν την πολιτική λιτότητας. Και αυτό διότι ήμασταν ειλικρινείς με τους πολίτες. Πιστεύω ότι αυτή η ειλικρινή αντιμετώπιση θα πρέπει να συνεχιστεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδυναμώνονται οι πολιτικοί, αλλά αντίθετα, πάρτε σαν παράδειγμα τη χώρα μας, ενισχύονται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ το λόγο εκ μέρους του κ. Βόλφμαν ε, σκεώδους για την πρόληψη και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών που συμμετέχει και στην Επιτροπή τη Διακοινοβουλευτική και του Ουσμπεκιστάν. Οι δέσμοι για την ε, οικονομική διακυβέρνηση και η διόρθωση των μακρονομικών ε, ανισορροπιών είναι ένα μέρος του όλου πακέτου ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και του χρέους. Οι ανισορροπίες είναι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και ε, χρήζουν μακροοικονομικής εποπτείας και στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξης. Ε, εάν υπάρχουν μακροοικονομικοί κίνδυνοι, πρέπει να παρακολουθούνται και να εντοπίζονται εγκαίρως εντός του πλαισίου που έχουμε ορίσει. Οι ανισορροπίες πρέπει να ε, εκτιμώνται και να αποτιμώνται με τα κατάλληλα εργαλεία, προκειμένου να υπάρχουν μηχανισμοί και δείκτες ώστε να καθορίζονται οι ανισορροπίες που προκύπτουν σε διαφορετικά τμήματα της οικονομίας. Οι διαδικασίες που προτείνει η Επιτροπή θα επιτρέψουν τα διαφορετικά μέτρα τα διερθωτικά μέτρα των κατώμελων συγγνώμη, και θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να δρουν και προληπτικά προκειμένου να αναχαιτίζουν αυτές τις ανισορροπίες αλλά και να έχουν την απαραίτητη προσαρμογή που έπειτα χρειάζεται. περιμένω την έκβαση της έκθεσης της κυρίας Φερέιρα, καθώς και τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων συναδέλφων, σκιωδών και εισηγητών, ώστε να δούμε και το διορθωτικό τμήμα της ε, μακροοικονομικής διακυβέρνησης. Thank uh, have... Ευχαριστούμε. κυρία Χούμπναρ. Ευχαριστώ. Και εγώ πιστεύω ότι η δέσμη αυτή είναι πολύ σωστή και θα πρέπει να προστατεύσουμε την, το περιεχόμενο. Οι κυρώσεις είναι ένα σημείο αφετηρίας για μας στην Ευρωζώνη. Θα έχουμε πάντοτε αυτή την ετερογένεια που παρουσιάζεται μεταξύ των μελών. Πρέπει να υπογραμμίσουμε και τα αίτια των ε, ανισορροπιών, ανταγωνιστικότητα ας πούμε. Αυτά θα συνεχίσουν να ισχύουν και στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν τα αίτια αυτά να τα έχουμε πάντοτε υπόψη και η οικονομική διακυβέρνηση να μην παραμένει αδύναμη γιατί θα πρέπει να παρακολουθεί και τις εξελίξεις και να προσαρμόζεται. Χρειάζεται λοιπόν προστασία και χρειάζεται να έχουμε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία θα είναι μια διαδικασία μάθησης. Θέλω να επικεντρωθώ τώρα σε δύο σημεία για τα οποία και εγώ ήδη έχω κάποιες αμφιβολίες. Νομίζω ότι ιδανικά θα χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να μην προκαλεί ανισορροπίες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό, αλλά η επιλογή μας σήμερα είναι να θεσπίσουμε ένα μηχανισμό, τον καλύτερο δυνατό, ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε όταν χρειάζεται στο επίπεδο της οικονομικής διακυβέρνησης για να διορθώνουμε τις κυβερνητικές πολιτικές. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη, σχεδιάζοντας αυτό το μηχανισμό, ότι θα χρειαστεί να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός συστήματος που να μην είναι τόσο επιρρεπές στις ανισορροπίες που σήμερα παρατηρούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα είναι άκρος χρήσιμο κατά το σχεδιασμό του συστήματος να μην διαχωρίσουμε τελείως τις εξωτερικές από τις εσωτερικές ανισορροπίες. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε το διτό χαρακτήρα των ανισορροπιών και άλλου συσχετισμού του, καθώ και το δίλημα μεταξύ τη ενοποίηση κάποιων πολιτικών και τη ανάπτυξη. Κάποιε φορέ το σωσίγιο μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ανισορροπιών ίσω να φέρνει λύσει, ίσω να πρέπει να ληφθεί μεταξύ των κριτηρίων που θέλουμε να καταγράψουμε. Επίση, χρήσιμο θα ήταν να θυμόμαστε διαρκώ ότι η Ευρωζώνη δεν είναι απλώ ένα σύνολο ε, μέρους κρατών μελών. Δεν αρκεί να παρατηρήσουμε δηλαδή την ατυνομική συμπεριφορά του καθενός. Όταν διορθώσουμε τις, ε, τις δυσλειτουργίες, όταν διορθώσουμε τις συμπεριφορές που δεν μας αρέσουν, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις επιπτώσεις που έχει η συμπεριφορά του καθενός στους υπόλοιπους στην Ευρωζώνη. Πιστεύω πάντως ότι τα μέτρα επιβολή που θα είναι το τελευταίο τμήμα του πακέτου του, της δέσμης και το τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά, όλο αυτό θα εξαρτηθεί από το σχεδιασμό του αρχιτεκτονήματος. Ε, εάν θα έχουμε κατανοήσει παρκώς ποιε είναι οι ανισορροπίε και ποια τα κριτήρια, πώς θα επιλέξουμε δηλαδή τους δείκτες, πώς θα τους συνδυάσουμε και πώ θα αξιοποιήσουμε τα στατιστικά μα δεδομένα. Θα πρέπει λοιπόν τα μέτρα αυτά βολής να ε, τα έχουμε διαρκώς κατά νου κατά το σχεδιασμό του τελικού συστήματος και για τις κυρώσεις το άρθρο 4 και τον κανονισμό περί μέτρων επιβολής. Εδώ κάπως παραξενεύομαι το, ως προς το πώς θα δικαιολογήσουμε τη λύση που θα προτείνουμε. Εδώ η ψηφοφορία μας έχει και πολιτικό χαρακτήρα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που εμπλέκονται για τις αντικειμενικές αξίες αναφοράς και το αν παραβιάζονται ή όχι. Ε, προσπαθώ να καταλάβω την όλη συλλογιστική, όμως νομίζω ότι εδώ καθοριστικός είναι ο ορισμός των εξαιρετικών, των εκτάκτων περιστάσεων. Στο παρελθόν όλοι είχαμε εμπειρίες από τέτοιους ορισμούς που δεν ήταν αρκετά καλά σχεδιασμένοι και προκαλούσαν τελικά βλάβες. Κάποιε φορέ βρισκόμαστε ανυπεράσπιστοι όταν προκύπτουν οι καταστάσει στην πραγματικότητα. Και το άλλο που θα πρέπει να μα να μας απασχολήσει κατά τις κυρώσεις στο άρθρο 4 είναι η έμεση ηθική βλάβη. Διότι τα κράτη-μέλη κάποιες φορές λέγεται ότι όταν δεν υπάρχει διαπιστωμένη παραβίαση θα εξετάσουν το κατά πόσο υπάρχουν παραβιάσει των αξιών αναφορά, θα συλλέξουν τα πρόστιμα και θα τα ανακατανείμουν μεταξύ του. Αυτό είναι κάπω περίεργο. Εφόσον είμαστε τόσο ευαίσθητοι στο ε, νηθική βλάβη, πρέπει να δούμε ακριβώ τι διαστάσει θα πάρει αυτό το θέμα στο Συμβούλιο και τι θα πυροδοτήσει ω προ τι κυρώσει. Για μένα δεν είναι ακόμη σαφέ. Ευχαριστώ, ο κύριο Γκίγκολτ. Πολύ σύντομα για τη δέσμευτη νομίζω η Επιτροπή έχει αναλάβει μια σοβαρή ευθύνη και πρέπει να θέσει σωστά τους οικονομικούς όρους του όλου θέματος. Η όλη συζήτηση στο Συμβούλιο δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να μας ικανοποιεί ως προς αυτή την άποψη. Όμως, ούτε και εδώ μπορούμε να δούμε το θέμα μόνον από πολιτικής σκοπιάς. Πρέπει να ξεπεράσουμε τις θέσεις που αναλάμβανε στο παρελθόν οι διάφορες πολιτικές παρατάξεις. Ξεκινάμε με την όλη συζήτηση βέβαια για τις κυρώσεις, καθώς και για το σύστημα επίλυσης, αλλά και τη διόρθωση των ανισορροπιών. Το σημείο φετηρία για τη δέσμη αυτή θα πρέπει να είναι οι πραγματικές ανάγκες για ισχυρότερη οικονομική συνεργασία και συντονισμό, βασιζόμενοι στις εμπειρίες που είχαμε από την πρόσφατη κρίση. Δεν καταπολέμουμε λοιπόν ανισορροπίες που είτε υπάρχουν είτε όχι, αλλά που έχουν πραγματικά επισημεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα στοιχεία αυτά που θα μας επιτρέψουν συνένεση, ε, να καταλήξουμε σε συνένεση, ώστε οι νέοι κανόνες να είναι συνολικοί και να απεικονίζουν τα διδάγματα που κομίσαμε από την πρόσφατη κρίση. Θα πρέπει να είναι και υποχρεωτικοί οι νέοι κανόνε. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει για τις, και για τι δύο πλευρέ. Και για το χρέο και το έλλειμμα από τη μια και για τι ανασορροπίε από την άλλη. Στι περιπτώσει όπου οι μεγαλύτερε οικονομίε στην Ευρωζώνη ουσιαστικά λειτουργούν αποπληθωριστικά, ενώ άλλοι έχουν ε, πολύ υψηλό επίπεδο πληθωρισμού, ε, όλο αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Και το μόνο πρόβλημα δεν είναι η ανταγωνιστικότητα. Έχουμε δικές και φούσκε με τις ε, τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και στην ανταγωνιστικότητα στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και τα μέτρα σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι σκληρά και αυστηρά. Υπάρχει περίπτωση να πετύχουμε ευρεία συνένεση μόνο εάν οι κανόνε είναι σκληροί και για τι δύο πλευρέ. Τι δύο όψει αυτών των προβλημάτων που έχουν συμβεί. Ε, Επίση, είναι σημαντικό να μην απαιτούμε από τι χώρε μετραλιτότητα τα οποία θα οδηγήσουν σε εξελίξεις αποπληθωριστικές Υπάρχουν και επιτυχημένες πολιτικές λιτότητας, όπου όπως είδαμε να συμβαίνει στη Σουηδία, που ξεκαθάρισαν ε, τα στραβά που υπήρχαν στη χώρα. Και μπορεί κανείς να υποφεληθεί από ισχυρότερε εξαγωγές, όπως έγινε εκεί, χρησιμοποιώντας ε, το ισοζύγιο και καλύπτοντας ε, την έλλειψη εσωτερικής ζήτησης που προκλήθηκε από τη λιτότητα. Αυτό όμως δεν ξέρουμε κατά πόσον μπορεί να το καταφέρει η Ευρώπη. Πόσε χώρε έχουν ξεπεράσει το όριο του 60% και θα φτάσουν το 80%. Εκεί θα υπάρξουν παρόμοιες αποπληθωριστικές τάσει, εάν δεν έχουμε ορθούς κανόνες. Δεν επιχειρηματολογώ λοιπόν υπέρ υψηλών επιπέδων δημοσίου χρέου, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε σωστά οικονομικά θεμέλια στις όλες μας προτάσεις. Διότι όλες οι ωραίες πολιτικές απόψεις εδώ θα μας οδηγήσουν σε βαθιά οικονομικά προβλήματα. Και η τελευταία παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι το ερώτημα το αν οι πιστωτέ θα πρέπει να εξαγοράζονται, να, εξαγοράζουν, να σώζονται από τα κράτη. Θα πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη εδώ ότι η αλλαγή της συνθήκης μπορεί να μην φέρει ακόμη αλλαγές στην πράξη, οπότε το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαγράψει δυνατότητες και προτάσεις για το πώς θα επιτυχάνεται ο στόχος αυτός χωρίς καμία ε, ε, προσαρμογή τη συνθήκη. Αυτό μπορεί να γίνει με κοινού κανόνε για τα κρατικά λόγου χάρη ομόλογα. Εάν το περιλάβουμε αυτό στου κανόνε των ομολόγων, των μελλοντικών κρατικών ομολόγων. Μπορεί να έχουμε ένα σύστημα λύση, μια προσέγγιση resolution scheme, χωρί να χρειάζεται και προσαρμογή τη συνθήκη. Υπάρχουν βεβαίω και άλλε δυνατότητε για να επιτευχθεί ο ίδιο στόχο. Όμω νομίζω ότι θα είναι υποδομητική αυτή η λύση. Είναι κάτι που μπορούμε να το προτείνουμε εμεί ω κοινοβούλια, γιατί και θα προασπίσουμε τα συμφέροντα των φορολογουμένων και δεν θα διασώζονται αυτοί που εύκολα πήραν πιστώσει από τι κυβερνήσει και τελικά θα καλύπτεται ο κίνδυνος που ανέλαβαν. Κυρία Σουίνμπεν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι έγιναν πολλά σχόλια Η δίκη θα περιοριστώ λοιπόν σε δύο σχόλια επί της διαδικασίας και δεν θα κάνω συγκεκριμένα σχόλια τα οποία θα τα κάνω με τους εισηγητές αργότερα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ισχυρότερη συνεργασία και το συντονισμό που αναφέρονται όλοι. Ε, θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως και δεν θα πρέπει να περιμένουν να γίνουν προτάσεις ε, νομοθεσίες. Πολλές από τις δράσεις θα μπορούσαν ήδη να αρχίσουν και νομίζω όσο πιο συντενισμένα είναι τα πράγματα, καλό θα ήταν να γίνουν όλα αυτά πριν, ε, πριν ε, περατωθεί όλη η διαδικασία. Και αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο να βρούμε το σωστό τρόπο, να μην γίνει γρήγορα απλώς και μόνον. Ε, ελάχιστες χώρες αυτή τη στιγμή τηρούν ε, τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ουσιαστικά δεν έχει σημασία γιατί οι κυρώσεις δεν θα αλλάξουν την κατάσταση για τα περισσότερα κράτη. Οι κυρώσεις ε, ούτως ή άλλως έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέτρα πρόληψης. Επομένως ε, θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα όταν θα έχουμε ισορροπία. Αν βιαστούμε δεν θα έχουμε αποτέλεσμα ε, πρέπει να έχουμε τις σωστές λύσεις ακριβώς επειδή υπάρχουν τεράστια δημόσια χρέη και επειδή υπάρχει πρόβλημα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σωστά και να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες ως συνήθως και να έχουμε μια καλή δημόσια κρέωση επί του σέματος, ε, διότι θα είναι η δυνατότητα που θα έχει το ευρύ κοινό να ακούσει τι ακριβώς συζητάτε. δεν θα πρέπει να έχουμε συμπληρωματικέ εκθέσει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ανοιχτά στι διαδικασίε μα και όταν θα φτάσουμε στο τριμερή διάλογο θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε συζητήσει όλα τα θέματα. Κάποια από αυτά είναι περίπλοκα οικονομικά θέματα και θα πρέπει να υπάρχει όλη η υποστήριξη που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μα για να μπορέσουμε να συντάξουμε αυτέ τι εκθέσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε σε ένα scoreboard ε, οικονομικών και χρηματοπιστωτικών δικτών και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη αυτών των δικτών. Τα κράτη-μέλη, ακριβώς λόγω του ε, τι συμβαίνει, ενδιαφέρονται το καθένα ατομικά για τα θέματα αυτά και τα, ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε ίσως να παίξει το ρόλο του διαιτητή. ίσως τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη ε, να επιβάλλουν την άποψή τους και κάποια μικρότερα κράτη-μέλη να βασίζονται σε εμά για να τα υποστηρίξουμε. Θα σταθώ εδώ για τα σχόλια και θα κάνω και μεμονωμένα σχόλια στους ε, εισηγητές. Ο κύριος Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι κάποια από αυτά που ακούστηκαν δεν ε, πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Μέχρι τώρα έχουμε το Σύμφωνο Ανάπτυξης και σταθερότητα, οι οποίοι αυτόματα προβλέπουν κάποιες κυρώσεις. Ε, αν κάτι δηλαδή δεν πάει καλά, υπάρχει αυτόματα η κύρωση. Αν κάτι πάει καλά, αντίθετα δεν προβλέπεται τίποτα. Οι συνέπειες αυτών των κυρώσεων είναι πάντα, όπως βλέπετε, η ανεργία. Οι συνέπειες ε, και η λογική, αν θέλετε, αυτής της πολιτικής είναι μια λογική την οποία επομίζονται οι εργαζόμενοι. Ήρθε λοιπόν και η κρίση και αυτό που εδώ ζητάμε είναι κυρώσεις. Κυρώσεις όμως με περισσότερη ευελιξία. Δεν αλλάζει τίποτα στον γενικότερο χαρακτήρα αυτής της πολιτικής. Δηλαδή, αυτό που ζητάμε είναι ένα σύστημα ποινικών κυρώσεων. Αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά ήταν ένοχοι τέτοιων ατασταλιών, τους λέγαμε ότι δεν διαχειρίστηκαν σωστά κάποια κονδύλια και προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπο να τους σώσουμε. Τι έγινε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Ε, το μόνο κριτήριο ουσιαστικά είναι να αυξηθεί ο ανταγωνισμός, αυτό το υπέστησαν τα πιο αδύναμα κράτη-μέλη και θα πρέπει πραγματικά λιγάκι τους επόμενους μήνες να πλησιάσουμε οι μεν τους δε σε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε από τη μία την κυρία Γκουλάρ, τον κύριο Λάμπερτ. Δεν πιστεύω ότι έχουμε ακόμα πλησιάσει την κοινή λογική. Ελπίζω να το πλησιάσουμε όταν συζητήσουμε για το σύμφωνο σταθερότητας, απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής. Και αυτό το ποινικό δίκαιο, αυτές οι πολύ αυστηρές κυρώσεις δεν θα πρέπει απλώς ε, να μας απασχολήσουν, θα πρέπει να δούμε την κοινότητα αυτή των κρατών, να την στηρίξουμε ιδιαίτερα όταν κάποια πιο αδύναμα κράτη-μέλη εξαιτίας της πολιτικής των πιο δυνατών κρατών μελών είτε της πολιτικής και της δραστηριότητας των χρηματαγορών πλήττονται με αυτό τον τρόπο. Σας ευχαριστώ. Κύριος Χουντής. Στο κυρία Πρόεδρε. Θέλω να δηλώσω εκ μέρους της ΓΚΟΕ, και ο συνάδελφος πριν, ότι επί της αρχής, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε αναλάβει καμία από τις εκθέσεις και από τη σκιά εντό εισαγωγικών θα παρακολουθήσουμε όλη αυτή τη συζήτηση, θα συμβάλλουμε ούτως ώστε να ακουστεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως, όμως, όμως ελπίζω να υπάρχει ο χρόνος και η διάθεση να ακούσετε και τις, επί της ουσίας απόψεις μας. Και εδώ θέλω να σας πω κύριοι συνάδελφοι ότι σε αυτό το πακέτο της δέσμης οικονομικής διακυβέρνησης που έχει εκπονήσει η Επιτροπή και νομοθετικές πράξεις θα επεξεργαστούμε εμείς, ε, η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε αντίθετοι. Η Επιτροπή δεν κατάλαβε τίποτα από την κρίση. Αυτό που κατάλαβε είναι ότι χρειάζεται περισσότερη πειθαρχία, περισσότερη εποπτεία, περισσότερος έλεγχος. Με συνέπεια, ένα βασικό πρόβλημα που εμφανίζεται σήμερα είναι το πρόβλημα της ανάπτυξης. Και έχω παρατήρησα και σημερινούς συζητητές, παρατηρώ και τα κείμενα, βλέπω και στην Ελλάδα δημοσιονομική πειθαρχία, ελλείμματα, ελλείμματα και βλέπουμε για την ανάπτυξη. Πότε θα γίνει επιτέλους αυτή η ανάπτυξη. Αυτό που δεν κατάλαβε κατά την άποψή μας η Επιτροπή είναι ότι όλο αυτό οικοδομείται σε λάθος βάση. Και από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου κύριε συνάδελφοι, το να ζητάς πειθαρχία σε λάθος εντολή, σε λάθος κατεύθυνση είναι καταστροφικό. Αναφέρομαι και εγώ στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Γιατί δεν το εφήρμοσαν οι περισσότερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο οι αδύνατε, αλλά ακόμα και οι ισχυρέ για ένα διάστημα. Δεν μπορούσαν να το εφαρμόσουν. Ήταν καταστροφικό. Διέλυε το δημόσιο. Διέλυε το κοινωνικό κράτο. Αυξανόταν η ανεργία. Δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό. Είναι αντιαναπτυξιακό. Αν δεν αλλάξει το σύμφωνο σταθερότητα, η όποια πειθαρχία θα έχει αποτελέσματα, ενδεχομένω στα δημόσια οικονομικά, αλλά θα έχει σημαντικότατα κοινωνικά προβλήματα. Και επειδή αναφερθήκαμε σε πειθαρχία και ακούστηκε πάλι το θέμα τη Εστονία, είχαμε κάνει και σχετική συζήτηση. Πειθάρχησε η Εστονία. Μπήκε στην ΟΝΕ ναι, η Εστονία, τι κοινωνικέ πλευρέ τη υπόθεση δεν τι ψάχνουν. Μισθή λιτότητα έω πείνα στου δημοσίου υπαλλήλου και ανεργία 20%. Αν αυτή είναι η στόχευση τη πειθαρχία, τότε δεν μπορεί κανεί να συμφωνήσει. Και ποιο δεν μπορεί να συμφωνήσει, κατά τη γνώμη μου. Δεν πρέπει να συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δεύτερο σημείο που θέλω να σας πω. Πράγματι, μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση, παρακολουθώ την προσπάθεια να ακουστεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι της Κομισιόν, έναντι του Συμβουλίου. Φοβάμαι, κύριοι συνάδελφοι, ότι η μάχη θα είναι δύσκολη. Μέσα από αυτές, αυτές οι διαδικασίες, επιτρέψτε μου να πω, και τέτοια μέτρα που μοιάζουν ότι νοικοκυρεύουν τα πράγματα αλλά είναι αντικοινωνικά, δεν περνούν πάντα με δημοκρατικέ διαδικασίε. Και το θύμα δεν είναι μόνο ο Ευρωπαίος πολίτης, είναι και οι εκλεγμένοι θεσμοί μέσα στο οικοδόμημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ακούστηκε στην οικοδόμηση του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού στήριξη, ενώ το προέβλεπε ω μορφή διεθνή συμφωνία, διεθνού συμφωνία το 218. Στην Ελλάδα, λόγω των αυστηρών και όλων αυτών των μέτρων, δεν ακούγεται το Εθνικό Κοινοβούλιο. Και εμεί, ω αντιπροσωπευτικό θεσμό, θα ενισχύσουμε διαδικασίε που λέει προληπτικά θα ελέγχουμε του εθνικού προπολογισμού, δηλαδή τα εθνικά κοινοβούλια ουσιαστικά θα παρακολουθούν τις εντολές και θα τις εφαρμόσουν. Πού πάει η έννοια της αντιπροσωπευτικότητας και της πολιτικής ευθύνης. Βεβαίως χρειάζεται ένα πλαίσιο συντονισμού και κοινή δράση, αλλά προς άλλη κατεύθυνση. Θέλω λοιπόν να σας πω, αυτό το διαπιστώνει και η Επιτροπή και ε, να μου επιτρέψετε και την έκφραση, μην κάνουμε πως δεν βλέπουμε τι γίνεται στο θεσμικό επίπεδο. Όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει εκτός των άλλων για αλλαγή των συνθήκων σημαίνει ότι κάτι πρέπει, κάτι θέλουν να αλλάξουν και να αλλοιώσουν το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε περήφανοι. Δεν έχουμε υποστηρίξει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά αν θέλει αλλαγή, δεν θέλει προς την κατεύθυνση αυτή που φαίνεται ότι υποχρεώνονται από τα πράγματα προκειμένου να περάσουν αυτές τις συνθήκες. Αυτό το σημείο θα σας παρακαλούσα να μην το προσπεράσουμε, θα το βρούμε μπροστά μας. Φοβάμαι λοιπόν ότι σε αυτή τη μάχη ισχύω μέσα στου θεσμού, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε δυσμενή θέση. Με αυτή την έννοια επαναλαμβάνω τη θέση αρχή παρόλα αυτά, ότι εμεί θα υποστηρίξουμε την προσπάθεια να ενισχυθεί η δική μα θέση, παρότι διαφωνούμε επί τη ουσία. Με αυτή την έννοια, για ενιαία θέση, με τέτοιε λογικέ, θα σα παρακαλούσα, κύριοι συνάδελφοι, να μην μα υπολογίζετε για ενιαία θέση σε τέτοιε λογικέ. Για την υπεράσπιση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ναι. Σα ευχαριστώ. Thank you, Mr. Euh, Αν μπορούμε να βρούμε μια λογική συνέπεια, ένα μάθημα από αυτή την κρίση, θα πρέπει να ξαναδούμε αυτές τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η Επιτροπή παραμένει στις διαπεριφερειακές ανισορροπίες των ελλημάτων και των εμπορικών συναλλαγών. Και φτάνει σε κάποια συμπεράσματα τα οποία θεωρώ ότι είναι αμφισβητήσιμα. Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες παραμένουν, αν θέλετε, μόνο το εμφανές τμήμα του iceberg. Υπάρχουν και άλλες ανισορροπίες που δεν τις εξετάζει η Επιτροπή. Πρώτον, η ανισορροπία μεταξύ αποταμίευσης και επενδύσεων στη Γαλλία και τη Γερμανία, π.χ δύο χώρες που ουσιαστικά είναι περίπου το 60% αυτών των ποσών, αυξάνονται οι Ευρωπαίες. Και την ίδια ώρα η αποταμίευση κάποιων τάξεων, των ανώτερων κοινωνικών τάξεων που αυξάνονται. Η Επιτροπή δυστυχώς με τις προτάσεις της απλώς επιδεινώνουν αυτές τις ε, ανισορροπίες κάνοντας πιο άκαμπτο το σύμφωνο σταθερότητας με περιοριστικές πολιτικές που δεν θα επιτρέψουν την ανάπτυξη να προχωρήσει. Ήδη είναι ευαίσθητη η ανάπτυξη. Δεύτερον, η προσαρμογή του κόστους των μισθών για να μην υπάρξουν ανισορροπίες στις, ε, εμπορικές συναλλαγές θα οδηγήσουν σε μία αποπληθωριστική πολιτική όσον αφορά τους μισθούς και τις αποδοχές. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν σημαντικά τα ελλείμματα. Οι κυρώσεις λοιπόν είτε είναι αυτόματες είτε είναι ή μη αυτόματες, δεν ξέρω τη διαφορά και αν υπάρχει ουσιώδης διαφορά, είναι δύσκολα να την καταλάβουν οι πολίτες μας. Θα πρέπει λοιπόν ε, το Κοινοβούλιο να στηρίχθει στην έκθεση πρωτοβουλίας του κυρίου Φεγιό που έδειξε την ανάγκη να δούμε τους δείκτες που αφορούν την επένδυση, την ανεργία, την ανάπτυξη και το ενδιαφέρον να εξετάσουμε την κάθε χώρα ξεχωριστά. Άλλο πράγμα η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία. Μια άλλη πάρα πολύ σημαντική έκθεση της κυρίας Μπέρες ε, για την κρίση. Τα συμπεράσματα της κυρίας Μπέρες δεν είναι αυτά στα οποία οδηγείται σήμερα η Επιτροπή. Και ο φίλος μου Γκίκολτ έκανε κάτι πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Το θέμα της ανισορροπίας ε, του εμπορικού ισοζυγίου σαφώς και θα πρέπει ε, να μας θέσει στην εξέταση του θέματος της χρηματοδότησης μέσω των κρατικών ομολόγων των διαρθρωτικών ταμείων. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να περάσουμε όλα αυτά τα θέματα και τις προτάσεις μας στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστούν τα εθνικά κοινοβούλια για την ορθότητα αυτών των προτάσεων. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να είμαι δυσάρεστη. Όμως, νομίζω ότι το βάρος που θα έχουμε ως Κοινοβούλιο έναντι του Συμβουλίου σε αυτή τη συζήτηση δεν θα εξαρτηθεί από την διάθεση των βουλευτών να δείξουν την πυγμή τους, αλλά να πείσουμε με την ποιότητα του έργου μας. Ποιότητα που αποδείξαμε και προς το Συμβούλιο και με τα κράτη-μέλη στα θέματα της εποπτείας. Ακριβώς γιατί οι βουλευτές που είχαν αναλάβει τα θέματα αυτά πήγαν στην ουσία των θεμάτων και κατήχαν τα θέματά τους πρότισαν, πρότειναν λύσει ε, ευρωπαϊκής εμβέλεια. Πιστεύω λοιπόν ότι και η δέσμη περί εποπτεία μας έδειξε ποια οδό πρέπει να ακολουθήσουμε και για την δέσμη που τώρα εξετάζουμε. Και το λέω ευθύ εξ αρχή, γιατί τίποτα εδώ δεν είναι αυτονόητο. Και ίσως εδώ να μην τους ευχαριστήσω όλους, αλλά θα πω ότι δεν έχω πίστη από την συζήτηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Οι εκθέσεις Φέγιο και Μπερές προκάλεσαν πολλά και αντιφατικά σχόλια. Διότι δεν έχουν ούτε ένα συγκεκριμένο σκελετό, ούτε συνέπεια. Εγώ καταλαβαίνω τη μέρημνα των εισηγητών να συγκεντρώσουν εδώ μία όσο το δυνατόν ευρύτερη πλειοψηφία. Όμως αυτή η συσπήρωση για μένα τουλάχιστον ε, αντικατοπτρίζει ένα πολύ βαρύ τίμημα. Δηλαδή, μη επιλογή η μη σωστή επιλογή μεταξύ πολιτικών και οικονομικών λύσεων. Μπορούμε λοιπόν την έκθεση αυτή να την ερμηνεύουμε ο καθένας όπως ε, θέλει. Πρέπει να πω ότι εγώ δεν θα συμφωνήσω με την κυρία Βόρτμαν Κόλ ότι ήδη το έργο έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό ίσα ίσα ε, το όλο θέμα για την οικονομική διακυβέρνηση που θα πρέπει να καλύψουμε μας υποχρεώνει να κάνουμε πολύ δύσκολες επιλογές. Και τις επιλογές αυτές πρέπει να τις κάνουμε για να ακουστεί η δική μας φωνή. Θα πρέπει να αποφασίσουμε αν είναι το Συμβούλιο ή η Επιτροπή που καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στη διακυβέρνηση της ε, Ευρωζώνης, της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Επίσης, αν είμαστε υπέρ των κυρώσεων ή όχι εάν πρέπει να ε, ε, ε, πυροδοτούνται αυτομάτως ή όχι. Θα πρέπει να επιλέξουμε. Τώρα ακούγοντας κάποιους συναδέλφους εδώ, νομίζω ότι αυτές οι επιλογές θα μας χωρίσουν. Μου φαίνεται αναπόφευκτο. Και για να ευχαριστήσω λίγο την κυρία Γκουλάρ, να θυμίσω τα λόγια του Φρανσουά Μπαϊρού που ήταν σαν δασκαλός της ότι όταν κανείς ε, δεν σκέφτεται κάτι δεν σκέφτεται τίποτα. Τέλο πάντων, η ουσία είναι ότι οι συγκεκριτέ πρέπει να θέσουν τα σωστά ερωτήματα επί τη ουσία. Ο ρόλο που έχουμε αναλάβει εδώ δεν είναι εύκολο, διότι το να έχουμε μια συνένεση βιτρίνα δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Δεν βρίσκω λοιπόν άλλη λύση από το να πω ότι θα πρέπει να εργαστούν σκληρά οι Ευρωβουλευτές που έχουν αναλάβει τα θέματα αυτά και ότι είναι τεράστιο το, τεράστια η πρόκληση που έχουν αναλάβει. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω σαν ε, πολίτης εκτός Ευρωζώνης. Η άποψή μου, εάν θέλουμε να διευρύνουμε την Ευρωζώνη, είναι ουσιαστικές ε, αυτές οι προτάσεις. Πρέπει να είναι αυστηρές, να έχουν συνέπεια, αλλιώς εγώ δεν πρόκειται να μπορέσω να πείσω τους πολίτες ε, της χώρας μου να ταχθούν υπέρ του ευρώ. Αυτό που λέμε εδώ είναι ότι αυτό που είπαμε το 2003 θα αποτύχει. Ότι οι χώρες αυτές δεν τηρούν τους κανόνες. Και τι έγινε, ακριβώς αυτό που είχαμε προβλέψει. Και νομίζω ότι ακριβώς την ίδια συζήτηση έχουν και στη Φιλανδία. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα κυρώσεων, τιμωρίας, όχι. Είναι θέμα να τηρηθούν οι κανόνες, πάκτα sunt servanda. Και καμία χώρα, μικρή ή μεγάλη χώρα, δεν πρέπει να παρεκκλίνει από αυτήν την δέσμευση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω γιατί δεχτήκατε μια προσθήκη στην έκθεση ΦΕΓΙΟ, ότι δηλαδή μπορούν χώρες ε, εκτός ε, να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαπραγμάτευση, εκτός ευρώ. Δεν θέλουμε τις χώρες αυτές ε, να προσχωρήσουν. Έχετε όμως εδώ κάνει ένα σφάλμα, διότι οι χώρες εκτός Ευρωζώνης σήμερα έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τις χώρες εντός. Και αυτό που είπε ο κύριος Γκίγκλ έχει δίκιο. Υπήρξαν κρίσεις στις χώρες αυτές. Προσπαθήσαμε να πειθαρχήσουμε. Κοιτάξτε τι έγινε με την Λετωνία. Αν τηρήσει κάποιος τους κανόνες, αν υπάρχει διάλογος ε, με τους πολίτες, θα επανεκλεγείται. Και πραγματικά δεν λέμε εδώ ότι η σταθερότητα είναι κάτι το αρνητικό. Είναι κάτι καλό για την δημιουργία ναι, αναπασχόλησης. Ο πληθωρισμός είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες μας. Σκεφτείτε μας λοιπόν, είμαστε απ' έξω και να είστε πιο ανοιχτοί. Ευχαριστώ. Το καλύτερο ήρθε στο τέλος. Όλοι οι συγητές, εάν επιθυμούν, έχουν ένα λεπτό για να απαντήσουν. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων βεβαίως. Μπορείτε αν θέλετε να πάρετε το λόγο και αργότερα με τους σκιώδες. Κυρία Βόρτμαν Κόλ. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την συνεισφορά τους στη συζήτηση. Βέβαια δεν είναι εύκολη η συζήτηση. Συμφωνώ με όλους αυτούς που είπαν ότι η έκθεση Φέιο και Μπέρες βασίστηκε σε συμβιβασμού. Εδώ πρέπει να μπούμε στην ουσία της νομοθετική μα εργασία, άρα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Γι' αυτό και ξέρω ότι η εργασία θα είναι δύσκολη, αλλά θα πρέπει να κινηθούμε, να υποχωρήσουμε σε ορισμένα σημεία όλοι μας, αλλά μόνο έχοντας μια ενιαία θέση με μεγάλη πλειοψηφία είμαστε ισχυροί. Θα πρέπει λοιπόν να υποχωρήσουμε, να δώσουμε και να πάρουμε σε αυτή τη συζήτηση. Θέλουμε να μειωθούν τα ελλείμματα και το χρέος. Θέλουμε να μειωθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτοί είναι οι δύο στόχοι μας. Ζητώ λοιπόν από όλους τους συναδέλφους που έχουν παρατηρήσεις, που έχουν συστάσεις, να έρθουν σε επαφή μαζί μου με τους άλλους συζητητές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα. Για την ενότητα, ναι. Ε, ευχαριστούμε, Αστρίτ, που είπες ότι δεν θα είναι απλό. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια. Και έπειτα, δουλειά, ναι, πρέπει να εργαστούμε σκληρά για τα θέματα αυτά. Δεν θα είναι απλό για κανένα από τα ζητήματα, για τα περισσότερα σίγουρα, και ευχαριστώ όσους μίλησαν για τα μέτρα τα σχετικά με τους κύκλους τους οικονομικούς, για όλη τη σύνεση που πρέπει να επιδείξουμε, για το ρυθμό που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι σωστό ότι πρέπει να είμαστε ε, ταχείς, πρέπει να δώσουμε ένα αποτέλεσμα ποιότητας. Και ε, εμείς ε, επίσης καταλαβαίνουμε την άποψη σας κύριε Σμίτ. Ευχαριστούμε κυρία Φόρτ. Ευχαριστώ. Ε, να θίξω κάποιες από τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ που αναφέρατε και τα καρότα και τα μπαστούνια. Πολύ σωστή υπενθύμηση. Και νομίζω ότι τα σχόλια περί ηθικής βλάβης ήταν πολύ πολύ σημαντικά. Αυτό είναι καθοριστική σημασία για τις κυρώσεις. Ε, είτε είναι αποτελεσματικές είτε όχι. Υπάρχουν τεράστια θέματα περί ηθικής βλάβης εδώ και σας ευχαριστώ και για τα δικά σας σχόλια γιατί θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ακριβώς να παρακάψουμε το ζήτημα της ηθικής βλάβης, κάτι που η Task Force, η ομάδα δράσης έχει αρχίσει να πράττει. Δεν είμαι βέβαιη ότι από την άποψη των επενδυτών η δική σας η λύση μπορεί να λειτουργήσει, γιατί για πολλούς από τους επενδυτές μας το θέμα είναι ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση λόγω του τραπεζικού συστήματος και των ομολόγων που αυτομάτως θα οδηγούν σε κάποιες εξορροπήσεις. Λοιπόν, ναι, να αναζητήσουμε λύσεις, αλλά σίγουρα αυτό θα το κοιτάξει και η ομάδα δράση. Και επειδή κοιτάμε όλα αυτά τα θέματα ως δέσμοι, είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να βασιστεί στο έργο που ήδη έχει γίνει. Όπω συζητούσαμε το πρωί και με του εισηγητές, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα μπορέσουμε να επωφεληθούμε από όσα ήδη υπάρχουν και εφόσον πάμε προς μια κατεύθυνση να δούμε τι μπορούμε να αντλήσουμε από τα ήδη υπάρχοντα για να επιτύχουμε το στόχο μας και να έχουμε αποτελεσματικές και λειτουργικές λύσεις για το μέλλον. Μάλιστα. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Να πω ότι στις 24-25 Ιανουαρίου θα έχουμε τις εκθέσεις. Έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και την υπομονή σας και που μπορέσαμε να διορθώσουμε αυτή την περίπλοκη συζήτηση σωστά. Και Απλώς να σας, ευχαριστώ, να σας ευχηθώ καλή όρεξη και θα τα ξαναπούμε στις 3 με τον κύριο Ταβάρες. Ευχαριστώ.